Welcome to the second part of our... Καλώς ήρθατε στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας σήμερα. Είχαμε μία μακρύτατη ψηφοφορία το πρωί. Πήραμε πολύ σημαντικές αποφάσεις. Θα περάσουμε στο σημείο 9 της μερίσιας διάταξης, ε, ε, περιορισμός των ανισοτήτων με ιδιαίτερη εστίαση ε, στην φτώχεια που πλήττει τα παιδιά. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια πρώτα απ' όλα θα μας μιλήσει για αυτό το ζήτημα που έχει ιδιαίτερη σημασία για την Επιτροπή μας ε, και για το Κοινοβούλιο. Η κυρία Τσούμπερ από την QNGL θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ μην υπερβείτε τα πέντε λεπτά. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλες τις οργανώσεις ε, που είναι σήμερα εδώ, Eurochild, ε, Eurochild UNICEF, Save the Children, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Φτώχειας και Solidar που δέχτηκαν την πρόσκληση της Επιτροπής μας στη σημερινή ακρόαση. Εμεί θεωρήσαμε ότι αντί να κάνουμε μια πρώτη σύσκεψη σκιωδών ήταν πιο ενδιαφέρον να ακούσουμε εκπροσώπου αυτών των οργανώσεων διότι έχουν στατιστικά στοιχεία για το θέμα αυτό και έτοιμες συστάσεις που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε στη σημερινή συνεδρία αλλά και στη μελλοντική συνεδρία με τους σκιώδεις εισηγητές για να δούμε ποιες είναι οι βασικές ιδέες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση που συντάσσω. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι για μένα ως Πορτογαλίδη είναι πάρα πολύ σημαντικό να συντάξω μια έκθεση με αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή στη χώρα μου γιατί εκεί γνωρίζω καλύτερα την κατάσταση ένα, από τα τρία, ένα στα τρία παιδιά πλήττονται από τη φτώχεια. Έχουμε συζητήσει με διάφορες οργανώσεις και από ό,τι φαίνεται το θέμα της παιδικής φτώχειας ε, δεν συνδέεται με ένα, μια ευρύτερη κοινωνική κατάσταση, ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε παρά να συνδέσουμε λοιπόν ε, την παιδική φτώχεια με τις ε, ελλείψεις κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας, παιδείας, με την ανεργία των νέων τις, με τις επισφαλείς θέσεις εργασίας ε, των ε, γονέων. Αυτές είναι οι βασικές αιτίες της ε, παιδικής φτώχειας. Οξύνεται δε αυτό το πρόβλημα σε πολλές χώρες προσλαμβάνει τραγικές διαστάσεις και οι εμπειρογνώμονες μας λένε ότι τα πρώτα θύματα της κρίσης και των μέτρων που επιλέχθηκαν για να αντιμετωπίσουμε την κρίση είναι ακριβώς τα παιδιά. Σε αυτή την προπαρασκευαστική εργασία που έκανα για την έκθεση, αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να συζητήσω με διάφορες οργανώσεις επιτόπου. Δεν νομίζω ότι είναι πρόσφορο να μιλήσω εγώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε καλύτερα τους εμπειρογνώμονες, αλλά να αναφέρω μόνο την περασμένη εβδομάδα ήμουν στο Σετούμπαλ στην Πορτογαλία και μίλησα με εκπροσώπους ε, μιας ε, οργάνωσης ενός ε, κοινωνικού βρεφονιπιακού σταθμού και βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότεροι γονείς παίρνουν το χαμηλότερο εισόδημα, το κοινωνικό μέρισμα ε, με 180 ευρώ το μήνα είναι όλο ένα και περισσότεροι οι γονείς αυτοί ε, που παρότι είναι καταρτισμένοι ε, χρειάζονται την στήριξη και όταν ζητούν και διατροφικό δελτίο πρέπει να αφαιρεθεί αυτό το ποσό από τα 180 ευρώ που παίρνουν μηνιαίως για το κοινωνικό μέρισμα. Πέρα λοιπόν από το υλικό πρόβλημα, τη φτώχεια, τα βασικά προβλήματα διατροφής, ε, ενοικίου, ε, στέγης, ε, υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα που διαγράφονται για το μέλλον, για την ε, πνευματική υγεία, για ε, τη, τους ψυχοκοινωνικούς ε, κινδύνους με τους οποίους βρίσκονται αντιμέτωποι αυτοί, αντιμέτωπα αυτά τα παιδιά βλέπουν από πολύ μικρή ηλικία σοβαρότατα προβλήματα στο σπίτι τους και δεν έχουν καμία δυνατότητα, καμία προοπτική για να φανταστούν ένα καλύτερο μέλλον. Μου είπαν στο βρεφονιβιακό σταθμό, λοιπόν, εκεί στο Σετούμπαλ, ότι τα παιδιά όταν παίζουν επιλέγουν σαν παιχνίδι να πούνε ότι α, θα πάμε στο ΝΟΕΔ. Όχι πάμε ξέρω εγώ, στο πάρκο ή ε, ε, να παίξουμε, γιατί αυτό ξέρουν ότι οι γονείς το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πηγαίνουν στο ΝΟΕΔ, να κάθονται στις ουρές για να βρουν ε, μία δουλειά. Και τα παιδιά παίζουν αυτό το παιχνίδι στο σταθμό. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν πρέπει να ε, τροποποιηθούν άρδιν οι πολιτικές που ακολουθούμε για να δοθεί μια απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν ε, να μην μακρηγορώ. Σας ευχαριστώ όλους ε, και προσβλέπουμε ανυπομονησία στη σημερινή ακρόαση. Σας ευχαριστούμε κυρία Τσούμπερ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους ομιλητές μας. Σας παρακαλώ να περιορίζεστε σε 5-6 λεπτά για τις παρεμβάσεις σας. Έτσι θα δοθεί ευκαιρία σε όλους να συμμετάσχουν. Η κυρία Χέινσουόρθ από το Eurochild θα αρχίσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μας δίνετε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στην ανταλλαγή απόψεων γιατί έδειξε αυτή η έκθεση για η δέσμευση του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσει η υπόθεση να προχωρήσει. Η κυρία Ζούμπερ ήδη τόνισε το βασικά το ότι ένα στα τρία παιδιά στην Πορτογαλία ίσως γίνονται αποκλεισμό και φτώχεια και ένα στα τέσσερα αντίστοιχα στην Ευρώπη. Και καταλαβαίνουμε ότι η παινία ε, κατά την ε, παιδική ηλικία έχει συνέπειες για όλη την ζωή. Οπότε το να μπορέσουμε να επενδύσουμε σε αυτό, δηλαδή στην πρόληψη αυτού του φαινομένου, αυτό είναι ε, κάτι το οποίο επιβάλλεται να γίνει από κοινωνική πλευρά αλλά και οικονομική, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην θεωρήσουμε το ζήτημα έχει απόλυτη πολιτική προτεραιότητα. Ε, ε, είμαστε το Eurochild. Έχουμε κάποιους φορείς που δουλεύουν με τα παιδιά και για τα παιδιά στην Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλά μέλη αλλά κυρίως προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες σε κάποια δίκτυα σε εθνικό επίπεδο, σε κάποιους ε, φορείς, σε συλλογικούς που προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά σε εθνικό επίπεδο. Ε, επίσης εκπροσωπώ εδώ και μια, ένα ευρύτερο συνασπισμό που λέτε EU Alliance for Events for Children, η Συμμαχία Ευρωπαϊκή για επενδύσεις για τα παιδιά και έχουμε εδώ πολλά 24 δίκτυα περίπου ε, συμμετέχει και η UNICEF τα χωριά και τα παιδιά αλλά επίσης για να καταπολεμηθεί η φτώχεια, η έλλειψη στέγης, η έλλειψη παιδείας και που θέλουμε επομένω αυτό που να καταφέρουμε είναι να μπορέσει να υλοποιηθεί η σύσταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2013 για επενδύσει χάρη των παιδιών, να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από πλευρά διηγημάτων των ανηλίκων και έτσι να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση. Οπότε μεγάλη μου χαρά ε, να εκμεταλλευτούμε τη σημερινή ευκαιρία, ούτω ώστε να δούμε τι θα γίνει και έχω εδώ πέρα αυτό το εγχειρίδιο ε, της εφαρμογής και υλοποίησης που το ετοίμασαν οι συντονιστές του Eurochild. Έχουμε 15 ε, μελέτες ε, για πολιτικές και πρακτικές που θεωρούμε ότι είναι οι βασικές αρχές όσον αφορά αυτήν την ε, σύσταση. Ελπίζουμε αυτό να εμπνεύσει αυτούς που χαράζουν τις πολιτικές ε, αυτούς όλοι που δίνουν τη μάχη για αυτή την υπόθεση γιατί η φτώχεια για τα παιδιά δεν είναι κάτι το μοιραίο είναι κάτι που εξαρτάται από τις πολιτικές ακόμα και όταν έχουμε σπάνιδα πόρων υπάρχουν επιλογές επομένως χρειαζόμαστε την πολιτική βούληση να δούμε τα πράγματα μακρόπνοα να επενδύσουμε εκεί που χρειάζεται και να εκμεταλλευτούμε ολονών τις δυνατότητες και αυτό τελικά θα αποδώσει Έχουμε επτά χαρακτηριστικά για την επιλογή αυτών των μελετών. Να σας πω τρία σχετικά. Πρώτα-πρώτα το ότι όλα αυτά δείχνουν ότι θα πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένη ε, αντιμετώπιση ε, επαγγελματική, να ξεπεραστούν κάποια μειονεκτήματα που δεν είναι θέμα επιδόσεων στο σχολείο, υγείας ή χρημάτων. Πάντα συνδυάζονται για αυτά τα φαινόμενα πολλοί παράγοντες. Άρα εδώ δεν είναι θέμα συντονισμό. Το θέμα είναι να υπάρχει διάλογο και διαφορετικέ προοπτικέ που να καταλάβουμε και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε κάποιες υπηρεσίε πρώτη γραμμή, σε επαγγελματίε που να δρούν επί τόπου, αλλά χρειάζονται υποδομέ. Γιατί έχουμε χάσει μεγάλε ευκαιρίε να μπορέσουμε να κάνουμε ήδη αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων και ιδίω αυτών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Επίση, ένα δεύτερο χαρακτηριστικό για μια καλή πρακτική είναι η ενεργή εμπλοκή των παιδιών και των οικογενειών τους. Είναι αδύνατον τα παιδιά να τα βγάλουμε από τη φτώχεια μόνο αν κάνουμε για αυτά ή και προς αυτά κάποιες ενέργειες. Βεβαίως και έχουμε θέματα διαρθρωτικά και αυτά τα φαινόμενα που τους ανθρώπους που αποκλείουν μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Μόνο από μέσα μπορούν να δοθούν οι λύσεις. Ε, και από μέσα θα παίξουν σημαντικό βέβαια. Χρειάζεται κάποιους επαγγελματίε να έχουμε που να υποστηρίζουν κάτι το οποίο κάνει μεγάλη διαφορά μακρόπνο. Οπότε και εμείς θεωρούμε ότι η πραγματική αλλαγή έχει σημασία όταν αυτοί που δημιουργούν την πολιτική και οι επικεφαλείς ε, θα καταλάβουν ότι έχει σημασία την υπόθεση και οπότε όπως τα είπε η κυρία Ζούμπερ είναι ότι δηλαδή θα πρέπει τα παιδιά να έχουν επίγνωση της αυτοτητά τους, το ότι μπορούν να έχουν θετικές σχέσεις με άλλους, ε, αυτογνωσία και τέλο πάντων να πάρουν τα ενία της ζωής τους στα χέρια τους. έτσι λοιπόν θα πρέπει να βλέπουμε και εμείς τα παιδιά στην κοινωνία μας. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι το ότι σε αυτό μας το δημοσίευμα βλέπουμε τι γίνεται και με την πολιτική και με την πρακτική. καινοτομία, επιχειρηματικότητα, να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Εντάξει, καλά είναι όλα αυτά. Αλλά χρειάζεται και μια δυναμική πολιτική που να καλύπτει τις επιμέρους ατομικές πρακτικές. Θα μιλήσουν γι' αυτό άλλοι συναδελφοί. Και εν κατακλείδη θέλω να σας πω συστάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτή σας την έκθεση. Πρώτα-πρώτα θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίως να συμφωνήσει με την προσέγγιση των τριών πυλώνων. Πρόσβαση δηλαδή σε υπηρεσίε και συμμετοχή των παιδιών όπω προτείνει η Κομισιόν. Ε, οπότε ε, θα πρέπει αυτό να το εγκρίνει το Συμβούλιο αλλά βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη ότι υπάρχουν περικόπες. Α, τρία, τρία, τρία. Α, δέκα, δέκα αυτά μας δώσατε. Οπότε να σα πω τι τρει παρατηρήσει μου και να κλείσουμε να προβάλλουμε το φαινόμενο αυτό στην μακροοικονομική θεματολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε να είναι ένας ε, δείκτης δεσμευτικός στον αφορά την ΟΝΕ, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εξωθηθούν, να έχουν υποστόχους της μακροοικονομικής πολιτικής να μειώσουν ε, την ε, μείωση και αυτό να μπήκε στο πρόγραμμα του Horizon 2020 και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αφιερώσει κάποιους ε, πόρους τόσο ώστε να παρακολουθήσει τη συνέχεια της πορείας αυτής της ε, σύστασης, δηλαδή την ευημερία των παιδιών, να παρακολουθήσει το πώς τα διορθωτική κατά μία χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της σύστασης στο ιστορικό των κρατών μελών. Και ποντάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι τώρα εισχαληθήκατε με τα δικαιώματα των παιδιών σε αυτή τη θητεία. Ο ρόλο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Αρχών, ε, το EEC, η εξωτερική υπηρεσία, τη... Ε, όλα, όλα τα θεσμικά όργανα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να βάλουν αυτό το θέμα σαν προτεραιότητα. Σας ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε την Εκατερίνα Τσέτσεγκ από την UNICEF. Ευχαριστώ. Εκπρόσωπο το ερευνητικό γραφείο της Φλωρεντίας της UNICEF. Ε, εκπροσωπούνται σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουμε μια ετήσια έκθεση ε, όπου βλέπουμε ε, τις επιπτώσεις της ύφεσης στα παιδιά. Βλέπουμε τις πλούσιες χώρες, χώρες που μέλη του ΩΣΑ ή κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αυξήσεις από το 2008 ως το 2012. Βλέπουμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις ε, στις χώρες όπου επλήγησαν περισσότερο από την χρηματοοικονομική ε, κρίση. Ελλάδα, Ισλανδία, Ιταλία, Ισπανία, τρεις βαλτικές χώρες, αλλά και η Ιρλανδία και Λουξεμβούργο. Και σε ορισμένο βαθμό και ε, χώρες όπως η Γαλλία και η Ουγγαρία. υπάρχει... 4,6 εκατομμύρια παιδιά περισσότερα που μετά την κρίση που πλήττονται από τη φτώχεια. Χρησιμοποιούμε το, για το 2008 το σχετικό ε, όριο αναφοράς ε, και ε, γίνεται προσαρμογή και στον πληθωρισμό. Δηλαδή συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Πρόκειται για παιδιά που βρίσκονται σε σε ομάδες, σε μεγάλες οικογένειες, παραδείγματο χάρη, ή με ε, οικογένειες μεταναστών, ή οικογένειες μακροχρόνια ανέργων. Επίσης βλέπουμε τις επιπτώσεις στους ε, ανέργους ε, βλέπουμε ότι για την ηλικία 15 έως 24 ε, έχει οξυνθεί το πρόβλημα κυρίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Επίσης αναλύουμε την επίπτωση της κρίσης ε, χρησιμοποιώντας ε, αντικειμενικούς δείκτες οικονομικής ευρωστίας και βλέπουμε ως προς το άγχος την ικανοποίηση ή την έλλειψη ικανοποίησης για τη ζωή, την ικανότητα να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται τα παιδιά, στον στον προβλημάτων στην ε, Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία αλλά και στην Τουρκία. Επίσης βλέπουμε ότι ε, από οικονομικής πλευράς έχουμε ε, πολύ αρνητικέ συνέπειες αλλά και εξαιρετικά ε, σοβαρές ε, κοινωνικές συνέπειες στα χαμηλόμιστα νοικοκυριά παραδείγματο χάρη και εκεί πέρα βλέπουμε και τη μεγαλύτερη αύξηση ανεργίας ούτως ή άλλως τέλος κλείνοντας εξετάσαμε τα επίπεδα δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα και παρότι αυξήθηκαν οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία κατά τη διάρκεια της κρίσης, ε, το ποσοστό των δαπανών που διοχετεύεται στα παιδιά και στις οικογένειες μειώνεται, ε, δηλαδή όταν χρειάζονταν ε, μεγαλύτερη προστασία δεν την έλαβαν και γι' αυτό ισχυριζόμαστε ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια προς τις οικογένειες και τα παιδιά σε περίοδους ύφεση θα πρέπει να είναι στον πυρήνα των απαντήσεων που δίνουν με τα παιδιά, διότι χρήζουν προστασία. ακόμη και αν δεν αυξήσουμε τις δαπάνες θα πρέπει να ε, διαχετεύουμε τα κονδύλια ευφιέστερα. Τέλος, το μήνυμα της UNICEF είναι να μην ξεχνάμε τα παιδιά ακόμη και σε χαλικούς οικονομικούς καιρούς και πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά ούτως ώστε όταν Ε, επέλθει η επόμενη κρίση δεν θα ε, παραμείνουν εξεχασμένα και θα έχουν κάποιο μέλλον. Αυτά και δεν θέλω να μακρηγορήσω κιόλα. Σας ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τώρα από την οργάνωση Save the Children την κυρία Σμολίνσκι. Καλώς σας απόγευμα. Ευχαριστώ για την οργάνωση της ανταλλαγής απόψεων για αυτή την πολύ επίκαιρη έκθεση για την παιδική φτώχεια. Ευχαριστώ επίσης που προσκαλέσατε την οργάνωσή μου. Σώστε τα παιδιά. Θα παρουσιάσω σύντομα την οργάνωσή μας, το έργο μας και την προσέγγισή μας στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας καθώς και κάποιες βασικές συστάσεις που έχουμε. Η οργάνωση Save the Children ιδρύθηκε το 1919. Η εργασία μας σήμερα βασίζεται στην εφαρμογή της συνθήκης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των παιδιών Έχουμε 13 ε, μάλλον εθνικές οργανώσεις στην Ευρώπη. Πέρσι τα μέλη μας ξεκίνησαν μια πανευρωπαϊκή έκθεση για τη φτώχεια των παιδιών και για τον κοινωνικό αποκλεισμό στην οποία έκθεση ξεκινήσαμε τη σύνταξή της δηλαδή έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε για τις επιπτώσεις της παιδικής φτώχειας αλλά και για να αλλάξουμε κάπως τις αντιλήψεις και να ζητήσουμε να εφαρμοστούν οι συστάσεις της ε, οργανωσής μας ε, ε, «Σώστε τα παιδιά». Βλέπουμε παιδική φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και σε αυτές έχουν υψηλό ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Άρα είναι πολιτική, είναι επιλογή η προστασία των παιδιών από την άποψη αυτή. Επομένως απαιτούνται και τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέτρα για να εφαρμοστούν οι πολιτικές αυτές. Στην έκθεσή μας γράφουμε επίσης ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση των παιδιών στη διάρκεια της κρίσης και βέβαια θίγει περισσότερο τα πιο ε, ευάλωτα παιδιά. Η φτώχεια των παιδιών είναι πολυδιάστατη. Πρώτα-πρώτα του στερεί την πρόσβαση σε δικαιώματα και ευκαιρίες. Μείωση εισοδήματος, που αυτό βέβαια καθορίζει αν ένα παιδί ζει σε φτώχεια ή όχι, από την άλλη μεριά μπορεί να μην αντιμετωπίζονται καν θεμελιώδεις ανάγκες των παιδιών όπως στέγη, ενδυμασία, τροφή κτλ. Επίσης οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό, σε αδυναμία πρόσβασης σε δομές όπως ε, παιδικούς σταθμούς κτλ. Επίσης και για την υγεία των παιδιών. Το ίδιο και για τον κοινωνικό αποκλεισμό που μπορεί να αποκλείσει τα παιδιά από κοινωνικές δραστηριότητες το, η οργάνωση «Σώστε τα παιδιά στη Φιλανδία» ξεκίνησε μια εκστρατεία την προηγούμενη εβδομάδα. Βρίσκουμε εκεί ότι παιδιά οικογενειών χαμηλών εισοδημάτων αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα χόμπι που έχουν ή άλλες ε, εξωσχολικέ δραστηριότητες και μάλιστα σε ορισμένες ε, περιπτώσεις υφίστανται και εκφοβισμό λόγω του χαμηλού εισοδήματο των οικογενειών τους. Τα αποτελέσματα, οι επιπτώσει μπορούν να είναι βαρύτατε λοιπόν για τα παιδιά. Ένα παιδί το οποίο περνάει από φτώχεια ένα χρόνο, ένα έτος δηλαδή, αυτό το νιώθει σαν ένα πάρα πολύ μακρότατο χρονικό διάστημα. Μερικά παιδιά μπορεί να μην μπορέσουν να αποκτήσουν τι απαραίτητε δεξιότητε που θα του επιτρέψουν να μπορέσουν με τη δουλειά του να ξεφύγουν κάποια στιγμή από τη φτώχεια. Η φτώχεια οδηγεί συχνά στην εγκατάλειψη του σχολείου, στην ε, νεανική ανεργία η οργάνωση Save the Children της Ισπανίας εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα έκθεση για το ίδιο θέμα, όπου αναλύονται σχολικοί και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ε, πρόσβαση των παιδιών στην ε, εκπαίδευση και βεβαίως και με τις αυξανόμενους ρυθμούς της φτώχειας στην ε, Ισπανία. Η πρόληψη τώρα της παιδικής φτώχειας πρέπει να βασιστεί στην εφαρμογή των σχετικών ε, συνθήκων. Το βλέπουμε και σε ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες ήδη εφαρμόζουν πολιτικές που ευθυγραμμίζονται με τη σύσταση αυτή της ε, οργάνωσής μας. Είναι λοιπόν ε, σημαντικό και αποτελεσματικό εργαλείο αυτό. Αλλά η εφαρμογή της στο εθνικό επίπεδο πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά. Και αυτό πρέπει να υποστηριχθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. επίσης ποιοτικές υπηρεσίες και οι οποίες να έχουν και οικονομικό χαρακτήρα, δηλαδή να είναι, να φθηνές με άλλα λόγια, αυτό εξαρτάται βέβαια και αν θα επιτευχθούν από τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα υπέρ των παιδιών και των οικογενειών τους. Η επένδυση, οι επενδύσεις μάλλον στην Ευρώπη πρέπει να αρχίσουν από τις επενδύσεις για τα παιδιά. Εκεί υπάρχει σημαντική προστιθέμενη αξία και αντιμετωπίζονται έτσι ταυτόχρονα πολλέ προκλήσει. Το νέο λοιπόν σχέδιο επενδύσεων θα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερε ευκαιρίε εάν συνδεθεί με επενδύσει στην κατάσταση των παιδιών. Περισσότερη φτώχεια και περισσότερο κοινωνικό αποκλεισμό τελικά θα σημάνουν βαρύτατο κόστο για τι κοινωνίε του μέλλοντο. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστούν και οι αιτίε τη φτώχεια του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, με προληπτική προσέγγιση όπως περιλαμβάνει η σύσταση επένδυση στο παιδί. Αυτή η επένδυση πρέπει να θεωρηθεί επένδυση και όχι κόστος. Έχω και την τελευταία μου διαφάνεια εδώ, αν έχετε την καλοσύνη να την εξετάσετε. Προβάζω εκεί τις βασικές μας συστάσεις προς τα ευρωπαϊκά όργανα. Πιστεύουμε δηλαδή ότι έχει έρθει η στιγμή να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα στην Ευρώπη και σε όλα τα παιδιά στην Ευρώπη. Θετικό μήνυμα που θα μπορούσε να είναι να εγκριθεί ο υποστόχος της Ευρωπαϊκής 2020 για τη μείωση της παιδικής φτώχειας. Επίσης, η εφαρμογή της σύστασης που ανέφερα πιο πριν πρέπει να είναι ορατή και να περιλαμβάνεται σε όλα τα σχετικά έγγραφα της Ένωσης. Και επίσης να εγκριθεί ένα, ένας οδικός χάρτης για την εφαρμογή της σύστασης επένδυσης στο παιδί. Να προβλεφθούν επίσης ειδικοί δείκτες για την παιδική φτώχεια και για τον κοινωνικό αποκλεισμό με στο το πλαίσιο της ε, σύστασης επένδυσης στο παιδί. Σημαντικό επίσης για μας είναι ακόμη οι δείκτες αυτοί να επιλεχθούν με ενεργό συμμετοχή των παιδιών και των νέων. Στην Ιταλία η οργάνωση ξεκίνησε ένα ίντεξ, ένα δείκτη δηλαδή που περιλαμβάνει και αυτούς τους δείκτες τους οποίους έχουν, στους οποίους έχουν καταλήξει με ενεργό συμμετοχή των νέων και των παιδιών. Τέλος δε, αλλά εξίσου σημαντικό, χρειάζεται μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα για την αντιμετώπιση της κοινωνικής στόχιας και η επένδυση στο παιδί θα πρέπει να αποτελέσει και έναν απόσπαστο μέρος του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ακολουθεί η κυρία Τζίλς από το European Anti-Poverty Network. Έχετε το λόγο κύριε μου. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε την Επιτροπή σας αλλά και την κυρία Ζούμπερ που μας εκάλεσε να μιλήσουμε στην σημερινή ακρόαση. Ταχείως, να σας πω ότι έχουμε με αυτό το δίκτυο κατά της ε, φτώχειας ένα εκτεταμένο δίκτυο με τις σχετικούς φορείς σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο 31 ε, δίκτυα από 18 φορείς. Προσπαθούμε να είμαστε ευγενείς προς εμάς, αλλά και εσείς θα πρέπει να ανταποδώσετε αυτή τη συμπεριφορά και στους άλλους ε, βουλευτές, αλλά και στους καλεσμένους μας. Ναι, αλλά ακόμη για το σημείο 8.2 δεν έχω λάβει Τη ε, τροπολογίες ακόμα. Στη σημεία που το είπαμε το πρωί. Τι να σας πω. Madam um, Καλώς. Οπότε είπαμε ότι πιστεύουμε στην συμμετοχή, θέλουμε να εμπλέκονται κάποιοι οι οποίοι έχουν ε, περάσει αυτή την εμπειρία της φτώχειας για να δούμε πώς θα εφαρμοστούν οι πολιτικές. Οπότε πιστεύουμε ότι από όλες τις φτώχειες η σημαντικότερη είναι η φτώχεια των παιδιών και προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται ε, και με την ε, συμπαράταξη με το Eurochild. Οπότε θεωρούμε ότι τώρα είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή γιατί όλο και αυξάνεται αυτή η φτώχεια. Ακούσατε τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά θα πρέπει να δούμε επίσης ποιες είναι οι τάσεις. Στα δύο τρίτα των κρατών μελών έχει αυξηθεί από το 2008 η φτώχεια των παιδιών. Θα πρέπει να δούμε ποιε είναι επίση οι αποκλήσει σε κάποιε χώρε όπω στην Ουγγαρία έχουμε 40%, στη Λετωνία 50%, Βουλγαρία, Ρουμανία επίση. Και αυτό ε, είναι δυναμή τη στα θεμέλια τη συνοχή στην Ευρώπη. Κίνδυνο επομένω, αλλά και ε, αυξημένε πιθανότητε κανεί να είναι στερημένο ω ενήλιξ. Οπότε βέβαια και η ανάπτυξη των παιδιών θίγεται έτσι και η υγεία τους. Αυτά είπε η κυρία Ζούμπερ καλά και επομένως ε, όλοι βγαίνουμε χαμένοι. Υπονομεύεται η συνοχή και αυξάνονται ε, οι δαπάνες, οι κοινωνικές, οι οικονομικές, μια από τα παιδιά δεν μπορούν ποτέ να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Και επομένως είναι θέμα επίσης και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε τα βασικά δικαιώματα, μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτό είναι θέμα κοινωνικό. Είναι μια χαμένη γενιά αθετούμε τις δεσμεύσεις μας προς αυτούς τους ανθρώπους. Είπαμε ότι τα φτωχά παιδιά μεγαλώνουν σε φτωχέ οικογένειε, αλλά να εξετάσει κανεί την φτώχεια των οικογενειών, αλλά δεν είναι δυνατόν κανεί να μην λάβει υπόψη ότι πρόκειται περί ατόμων που έχουν ατομικά δικαιώματα. Ε, μιλώ για του ανηλίκου. Οπότε θα πρέπει να δούμε την πρόοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα πλαίσιο πολιτική, έχουμε αυτήν την. Ε, σύσταση, αλλά δεν υλοποιείται. Δεν διαπιστώνουμε να υπάρχει προβολή αυτού του θέματος, να υπάρχει πολιτική ε, βούληση και επί τη βάση του πλάνου Juncker. Να δούμε τι θα γίνει με τον στόχο για το 2020, να δούμε να μην ε, χάσουμε ε, από την προσοχή μας τον στόχο αυτό στα πλαίσια του ορίζον. Επίσης να δούμε τι θα γίνει με τη συστημική προσέγγιση, να δούμε τις διορθωτικές αιτίες της φτώχειας των παιδιών, ανισότητα για την κατανομή των πόρων. Αυτό είναι πολύ βασικό για τη δημιουργία, τη γέννηση αυτής της φτώχειας. Οπότε κανείς, εάν αυτό το ξεχάσει, ε, εξετάζει ε, κατά περίπτωση λύσεις ούτε να ε, κατηγορούμε τι οικογένειε, γιατί πάλι θα καταλήξουμε σε εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Να δούμε την ανισότητα, να δούμε τις ε, ανισότητε και αποκλήσει των χωρών. Περίπου στα μισά κρατημέλη αυξάνονται οι ανισότητε. Και ε, ποιε είναι οι αιτίε, αυτά που τα έθιξε η κυρία Ζούμπερ. Είναι θέμα κατανομή. Τι γίνεται με το εισόδημα, τι γίνεται με του μισθού. Μιλάμε για το 8,9%. Το 1 τρίτον δε των φτωχών έχουν δουλειά. Πάνω από το 50% των ε, οικογενειών στη Βρετανία, των φτωχών, έχουν δουλειά. Αλλά τι θα γίνει, Και θα γίνει τα συστήματα κοινωνική προνοία. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κενό το οποίο δεν έρεται. Έχουν το 2013 μια έκθεση για τις ανισότητες και εκεί είδαμε ότι έπεσε το εισόδημα. Όμως τα φορολογικά συστήματα βοηθούσαν όλο ένα λιγότερο. Να πώς απέτυχαν τα κράτη να εξασφαλίσουν ε, την υποστήριξη των πιο των λιγότερο τέλο πάντων προνομιούχων μέσα από το σύστημα κοινωνική προνοία. Θα πρέπει επίση να δούμε ποιε είναι οι επιπτώσει τη κρίση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, από τη UNICEF και από το CDC κάποια στοιχεία. Επίση έχουμε και τον φόρο για τι καθολικέ υπηρεσίε. Πολύ σημαντικό αυτό για να δούμε πώς θα εστιατεί η προσοχή μας και να δούμε τι τελικά όσον αφορά το εισόδημα υπονομεύει τη θέση των παιδιών γιατί κάποια παιδιά κινούν περισσότερο από άλλα. Να, γιατί οι καθολικές υπηρεσίες είναι σημαντικές. Μιλούμε για μεγάλες οικογένειες, για μονογονικές οικογένειες, για άτομα σε δύσκολες καταστάσεις, μόνους ε, ε, μετανάστες, τους ε, Ρωμά με τις διακρίσεις και πάρα πολλοί πάνε να δουλέψουν αλλού, ας πούμε στη Λετωνία. Πολλοί γονεί πάνε να δουλέψουν σε άλλη χώρα και αφήνουν πίσω τα παιδιά. Να και ένα άλλο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα, όσον αφορά τι ε, συστάσει, ε, τι έχει μέχρι τελευταία στιγμή, πολιτική βούληση χρειάζεται για να μπορέσει αυτή η θεματολογία να προχωρήσει, για να, μην κάνουμε, για να κάνουμε κάτι για την ανισότητα, τη φτώχεια και τη φτώχεια των παιδιών, να γίνουν όλα αυτά στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Προτεραιότητε. Με συγκεκριμένε συστάσει θα θέλουμε να υλοποιηθεί ε, το, υπόθεση των ε, δικτών των επιδόσεων και έτσι επομένως να προχωρήσει η σύσταση για τις επενδύσεις για τα παιδιά, συστημική προσέγγιση για τις ανισότητες. Να δούμε πώς θα υπάρχει σε όλη τη ζωή κάποιο επαρκές εισόδημα. Ευρωπαϊκά στάνταρ για τους μισθούς που να είναι αξιοπρεπείς και οι μισθοί και το εισόδημα και οι εργασίες και το ελάχιστο εισόδημα. Άρα να δούμε τι γίνεται σε δύο μέτωπα. μισθού και δουλειέ και εισόδημα τέλο πάντων. Και έτσι να έχουμε προοδευτικό φορολογικό σύστημα στις καθολικές υπηρεσίες που να είναι προσβάσιμε και να υπάρχει επομένως ένα τέτοιο πλαίσιο και να έχουμε επομένω ολοκληρωμένη στήριξη για τις οικογένειες και τα παιδιά ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια των ανηλίκων. Επίση, παρακαλώ να πω ότι χρειάζεται συμμετοχή απευθύνω έκλεισε. Είναι σημαντικό να δούμε πώς οι νέοι και τα παιδιά μπορούν να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Και να μην κοιτάει ο καθένας την ατομικό του σταυρό. Ε, γιατί αν κάποιος ε, εμπλέκεται, κατόπιν τον ακούνε πιο προσεκτικά και ενωσιακά και σε εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε κυρία Τζόουνς. Ε, τώρα ο κύριος Κόνι Ρόιτερ από το Σολιντάρο, τελευταίος ομιλητής μας, θα πάρει τον λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ διότι είμαι και ο μόνος άντρας στο πάνελ αλλά δεν νομίζω ότι είναι γυναικείο αυτό το, το ζήτημα. Χαίρομαι που αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις βασικές αιτίες και πώς να βοηθήσουμε αυτούς που το χρειάζονται, περνώντας κάποια πολιτικά ζητήματα. Συγγνώμη, αλλά είμαι πολύ γρήγορος και πέρασα τη, προσπέρασα τη διαφάνεια. Ε, βλέπουμε μέλη της Solidarity που συμβάλλουν ε, στην καταπολέμηση της στόχης όπως η Solidarité Laïque στη Γαλλία και άλλες αντίστοιχε οργανώσεις στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει και μια άλλη από την Αυστρία διάφορες οργανώσεις ε, που δεν περιορίζονται στα λόγια αλλά επιτέπου δρούν διότι είναι πραγματικότητα παιδική φτώχεια και όχι μόνο στις χώρες της ύφεσης με ε, υπάρχουν ε, υποδειγματικές χώρες όπως η Γερμανία που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, είναι κοινωνικό το ζήτημα διότι είναι στο τέλος ε, της αλυσίδας η παιδική φτάχη αλλά τελικά οδηγεί σε απομόνωση και στις οικογένειες, στις φτωχές οικογένειες, οι γυναίκες και τα παιδιά είναι τα μεγαλύτερα θύματα. Πώς μπορεί κάποιος να δώσει μια απάντηση, οι κοινωνικές υπηρεσίες, παραδείγματο χάρη υπηρεσίες στον τομέα ε, της παιδείας, ε, της υγείας, ε, κοινωνικές υπηρεσίες, στέγη, εργατική στέγη, λύσεις, ούτως ώστε να ξεφύγουν από την παγίδα της φτώχειας τα παιδιά. Εάν συζητήσετε με ψυχολόγους θα δείτε ε, ότι ε, ακόμη και πριν να πάνε στο σχολείο, πριν τα έξι χρόνια τους, ε, αν βιώσουν κάτι τέτοιο τα παιδιά πολύ δύσκολα μπορεί να το ξεπεράσουν μελλοντικά. Πρόκειται λοιπόν για επένδυση στους ανθρώπους, όχι μόνο στα παιδιά, όπως μας είπε και η συνάδελφος από τη UNICEF. Είναι πολύ σημαντικές οι δυσκολίες, ε, διότι πρόκειται για τη σκληρότερη μορφή της φτώχειας. Εμείς αγωνιζόμαστε για την κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω. Και η Σολιντάρ προσεγγίζει το ζήτημα μέσα από την απασχόληση και τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη εσείς, η Επιτροπή Απασχόλησης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασχοληθήκατε με ζητήματα όπως η απόσπαση των εργαζομένων, ε, τις ε, μονοπρόσωπες εταιρείε περιορισμένης ευθύνης, ε, αλλά το θέμα, ένα εγκάρσιο ζήτημα είναι ποιες είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις στις οικογένειες και στα παιδιά όλων αυτών των ζητημάτων ε, και πώς επηρεάζεται η κατάσταση ε, στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Έχουμε φοβερά προγράμματα μηδενικών ορών, παραδείγματος χάρη ευέλικτες μορφές εργασίας και άλλα τέτοια μεγαλεπίβολα σχέδια. Βλέπουμε όμως ε, ότι μας απασχολούν και ζητήματα όπως συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ε, ζωής. Ε, όμως ξέρετε ότι η αγορά εργασίας είναι τέτοια που δεν υπάρχουν, υπάρχουν όλα είναι και λιγότερο δυνατότητες να συμφιλιώσει κανείς την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή προστατεύοντας και τα παιδιά. Οι επενδύσεις στον τομέα της παιδείας είναι ένας κοινό στόχος, φαντάζομαι, και σίγουρα το εξετάζετε και εσείς το ζήτημα, τι σημαίνει να κάνουμε πολύ ωραίες ομιλίες και να συμπεριλαμβάνουμε αυτά τα στοιχεία στην ότι χρειάζονται επενδύσεις, αλλά τελικά λέμε ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και τα κράτη-μέλη δεν διοχετεύουν τα απαιτούμενα κονδύλια και δεν τα έχουν κιόλα, διότι όταν μιλάμε για τη δημοσιονομική εξυγίανση, οι δαπάνε για την παιδεία θεωρούνται κόστο που πρέπει να περικοπεί και κανεί από πλευρά Τρόικα δεν συζητάει για τι κοινωνικέ επιπτώσει αυτών. Λένε όλοι πρέπει να καταπολεμήσουμε την παιδική φτώχεια. Ναι, πρέπει να αναχαιτιστεί η φτώχεια, αλλά τελικά οι πολιτικές έχουν αντίστροφα αποτελέσματα και ε, ε, αυτό έτσι καλλιεργείται σε έφορο έδαφος ο λαϊκισμός, η προπαγάνδα με τα γνωστά αποτελέσματα και την άνοδο της ακροδεξιάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε ε, μικρή ηλικία θα πρέπει να αρχίσει η δράση και να θεωρείται ως ένα απαιτούμενο βήμα να γίνονται οι κατάλληλες δημοσιονομικές επιλογές και να διοχετεύονται σωστά τα κονδύλια. Τα σχολικά μας συστήματα δεν μας επιτρέπουν πάντοτε πρόσβαση, καθολική πρόσβαση για όλα τα παιδιά. Ε, η καλύτερη επένδυση είναι να θεωρείται η παιδεία δημόσιο αγαθό. Μου έχουν μείνει δύο δευτερόλεπτα και ήθελα να αναφερθώ σε ένα εξίσου σημαντικό κατά πρόβλημα. Πέρα από την παιδική φτώχεια θα πρέπει να ασχοληθούμε και το θέμα των παιδιών των μεταναστών που ε, λειτουργούν, ε, διαβιούν παράνομα σε μια χώρα και δεν έχουν πρόσβαση στις στέγες, κοινωνικές υπηρεσίες και στην παιδεία. Καλωσορίζω από αυτού και ε, την έκθεση της Νάταλη Γκρίσπεκ, διότι όταν μιλάμε για την παιδική φτώχεια στην άκρη της αλυσίδας, καταλαβαίνετε ότι η φτώχεια των παιδιών μεταναστών είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα των ανισοτήτων που πλήττουν την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Η κυρία Μελάν είναι τώρα εγγεγραμμένη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πρώτα θέλω να επισημάνω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι να δείξουμε μια ταπεινότητα όταν μιλούμε για φτώχεια, ενώ όλοι μας εδώ έχουμε πολύ υψηλά εισοδήματα, καθώς το ίδιο και για την απασχόληση, ενώ είμαστε από τους πιο προνομιούχους της κοινωνίας. Κατά τα λοιπά, τα παιδιά για τα οποία μιλούμε είναι παιδιά τρίτης γενεάς πλέον της οικοδόμησης της Ευρώπης και της παγκοσμιοποίησης και είναι απολύτως τα θύματα αυτών των δύο κινήσεων. Γιατί? Διότι η παγκοσμιοποίηση αλλά και η οικοδόμηση της Ευρώπης ανέτρεψε όλα τα σημεία αναφοράς και ιδίω από δύο αιώνες έχει οδηγήσει σε μια επιστροφή στις αρχές του 19ου αιώνα με μια βαθύτατη φτώχεια απολύτως απαράδεκτη. Άτομα που βεβαίω είναι οι γονεί, δεν έχουν την ικανότητα να προσφέρουν στι οικογένειε τους αξιοπρεπείς συνθήκες διαβιώσεως. Και αυτό οφείλεται στην ανατροπή όλων των συστημάτων που είχαν θεσπιστεί μετά τους πολέμους, που ήταν φρικτοί, αλλά που μετά οδήγησαν στην οικοδόμηση της Ευρώπης και στην παγκοσμιοποίηση. Βέβαια και πρέπει να εγκύψουμε στις ε, έγνοιες των παιδιών και της φτώχειας, αλλά να μην κάνουμε λάθος. Δεν μπορούμε να ανακατεύουμε τα συμπτώματα με τα αίτια. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα και στις οικογένειες και στα κυρίαρχα κράτη την δυνατότητα κυρίαρχα να ρυθμίζουν τα των οικονομιών τους και όχι με άνωθεν επιβολή νόμων διότι εκεί καταλήγουμε, φτιάχνουμε θύματα. για να αποφύγουμε να έχουμε μια χαμένη γενιά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω για την μελέτη επένδυση στο παιδί. Και όπως λέχθηκε κιόλας στη μελέτη, νομίζω ότι η μελέτη έχει αξία. Μιλεί για τη σημασία στήριξης της παιδείας για τις μη προνομιούς ομάδες. Επιθυμώ να σχολιάσω αυτό που είπε η συναδελφός μου μόλις είπε ότι αρμόδιες είναι οι χώρες μέλη. Δεν νομίζω ωστόσο ότι οι χώρες μέλη είναι υπεύθυνε για τους... Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, η Τσεχία για παράδειγμα στήριξε πολλές φτωχές οικογένειες με υποστήριξη, με χρηματοδοτική υποστήριξη που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο ότι οι οικογένειες από μη προνομιούχα περιβάλλοντα έχουν ε, περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο. Αν στόχος είναι να συμπληρώνουν την δευτερεύουσα εκπαίδευση, φαίνεται καθαρά ωστόσο ότι οι παιδιά από φτωχές οικογένειες δεν μπορούν να τα καταφέρουν να τελειώσουν το σχολείο. Φτωχά παιδιά γίνονται και φτωχοί γονείς. Και ε, χρειάζονται συστήματα υποστήριξης, αλλά κυρίως το βάρος πρέπει να δοθεί στα συστήματα παιδείας. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φανεί καθαρά ότι τα συστήματα παιδείας επιτρέπουν να ξεπεραστούν κάποια όρια και για τα ε, φτωχά παιδιά, παιδιά από φτωχέ οικογένειε δηλαδή. Ποια είναι άραγε η λύση, με ποιο τρόπο μπορούν, μπορεί κανείς να βοηθήσει τα παιδιά στο σχολείο, τους μαθητές, τους σπουδαστέ, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να βρουν καλύτερες δουλειές στο μέλλον. Εγώ αναμένω με μεγάλη υπομονησία την έκθεση που τη βρίσκω πολύ σημαντική. Οι αρμοδιότητες ε, στην παιδεία είναι βεβαίως αρμοδιότητες που ανήκουν στην κάθε χώρα μέλος, αλλά μπορεί να δοθεί μια συνολική υποστήριξη προς τις χώρες μέλη. Ευχαριστώ, η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο ακούμε, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν 2015 έχουμε αύξηση της παιδικής φτώχειας και συμφωνώ ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε τις αιτίες, τα αποτελέσματα, τις αιτιώδεις σχέσεις τέλος Βλέπουμε ότι θα έπρεπε αυτό να είναι φαινόμενο τριτοκοσμικό. Όμως στην Ευρώπη αυξάνονται τα σχετικά αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε βέβαια την παγκοσμιοποίηση, έχουμε τον νεοφιλελευθερισμό, έχουμε την κυριαρχία των τραπεζών και των ε, πολυεθνικών, ε, τους ολιγάρχες, έχουμε όλο αυτό, τη διαπλοκή της διαφθοράς, όλα αυτά είναι στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτά είναι η αιτία της φτώχειας. Μιλώ για τη φτώχεια και των ενηλίκων και των παιδιών. Δεν ξέρω, υπάρχει εδώ κάποια διάκριση ε, τι, ε, τι έχουν να μας πούν οι εμπειρογνώμονές μας, να δούμε τι προσέγγιση είναι πιο δόκιμη για το πρόβλημα. Φυσικά και σε οικογένειες ε, μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά και πολλές φορές η, μόνο από μόνο από τη μητέρα οπότε και είναι πιο πολύ εκτεθειμένα στην φτώχεια. Αλλά πολλές φορές υπάρχει διαφορά μεταξύ πλήρους οικογένειας ή μονογονεϊκής. Θα πρέπει επομένω ε, να θυσιάσει κανεί τα πάντα για να θρέψει τα παιδιά, για να τα στείλει στο σχολείο και για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες τους. Επομένως η φτώχεια και των ενηλίκων και των ανηλίκων είναι φαινόμενα τα οποία έχουν κάποια επικάλυψη. Να δούμε τώρα επομένως πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα φαινόμενο και το άλλο. Τι διαχωρισμό υπάρχει στους τρόπους αντιμετώπιση. με φτωχού γονεί και στερημένα παιδιά δηλαδή. Ανέφερε τις, ε, ε, την Ουγγαρία κάποιος ομιλητής που είπε για τι ανισότητε και είπε ότι έχουμε 40% φτώχεια παιδιών στη χώρα μου και αυτό είναι συγκλονιστικό. Θα ήθελα να μάθω ποιε είναι οι πηγέ, αλλά ενδεχομένω είναι αληθέ. Οπότε πώ είναι δυνατόν μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 χρόνια έχει τέτοιους ρυθμούς ε, παιδικής φτώχειας. Τέτοια ποσοστά. Βεβαίω και είναι θέμα τι είδου επασχόληση υπάρχει, τι είδου μισθοί υπάρχουν. Πάντω, ε, ας πούμε, έχουμε κάποιους εργάτες βιομηχανικούς ε, και οι οποίοι έχουν ετήσιο μισθό 200-250 ευρώ. Έχουμε μια νοσοκόμα που παίρνει 350 ευρώ δουλεύοντας ε, τρεις διαδοχικές βάρδιες σε νοσοκομείο. Άρα τι να κάνουν οι Ούγγροι γονείς για να αποφύγουν αυτή την παινία των παιδιών. Θα πρέπει να κάτσουμε για να χτυπήσουν το κακό στη ρίζα του και να μην, να μην, ξε, χάνουμε τον προσανατολισμό της συζήτησης. Και χτες έγινε μια συζήτηση ε, και φόρουσε τους Ούγκρους γονείς και τους ρωτήσαμε ποια είναι η αιτία της δικής τους φτώχειας. Μα είπανε ότι είναι οι άδικες πρακτικές των τραπεζών. Επίσης τα μισθωτήρια που τους επιβλήθηκαν γιατί ε, επίσης κάποια δάνεια γιατί στην δεκαετία 2003-2013 είχαμε τριπλασιασμό των, ε, του, του, του, του ποσού αποπληρωμή του δανείου σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο. Άρα, άμα ρωτήσει κανείς κάποιους γονείς τι γίνεται, γιατί είναι φτωχοί. Θα του πει είναι φτωχοί γιατί του κλέψαν οι τράπεζε. Ε, άρα α κάτσει να σκεφτεί τη λύση από αυτή τη βάση Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις ε, των εκλεκτών προσκεκλημένων μας. Ε, είπαμε πάρα πολλά πράγματα για τις αιτίε της φτώχειας. Όταν ε, μιλάμε για τη φτώχεια δεν εννοούμε μόνο την ηλική διάσταση, τα χρήματα, διότι Εξίσου σημαντική είναι η έλλειψη παιδείας, στέγης και η βία συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής ε, βίας. 12χρονα ε, παιδιά ε, στη Σλοβακία εκπορνεύονται λόγω της φτώχειας. Στην ε, Σλοβακία είναι 12% το ποσοστό των παιδιών που απειλούνται από τη φτώχεια. Είναι υπερβολικά υψηλό το ποσοστό. Υπόθηκε ότι είναι εθνική αρμοδιότητα. Η απάντηση που μπορεί να δοθεί σε αυτό το πρόβλημα. Πάντως, ε, σε κάθε περίπτωση μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Θα πρέπει να βοηθηθεί ολόκληρη η οικογένεια και όχι μόνο ένα κομμάτι. Θα πρέπει να προσφέρουμε ποιοτικές ε, θέσεις εργασίας και υπηρεσίες στους γονείς. Και μιλώντας γι' αυτό, στη Σλοβακία παρατηρούνται προβλήματα ακόμη και με τον βασικό μισθό. Δηλαδή δεν δηλώνεται ολόκληρο το, ολόκληρη εργασία κάποιου, έτσι χάνονται ε, συντάξιμα δικαιώματα, διότι δηλώνεται μόνο ο βασικός μισθός και το υπόλοιπο πληρώνεται παράνομα. Αυτό στην περίπτωση που έχει κάποιος δουλειά. Είδαμε για την Τσεχία και για την ε, Σλοβακία κάποια στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι μετά ε, την ηλικία των δύο δεν υπάρχουν κρατικές υποδομές ε, φύλαξης των παιδιών για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των γονέων. Χρειάζεται στοχευμένη βοήθεια λοιπόν ένα επίδομα για τους γονείς. Βεβαίως όμως αυτό που συμβαίνει είναι ότι παίρνουν το επίδομα οι γονείς αλλά δεν ε, υποφελείται το παιδί και παραμένει μέσα στην ε, φτώχεια. Όταν ε, ένα παιδί προέρχεται από μη προνομιακό περιβάλλον, δύσκολα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και στην πράξη θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της παιδείας χωρίς αποκλεισμούς. Ε, αυτό σημαίνει ότι ανεξαρτήτως προέλευσης, ε, ε, περιβάλλοντος, κοινωνικής τάξης δεν θα υπάρχουν διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και πέρα από το σχολείο χρειάζεται ποιοτικό χρόνος για τα παιδιά στον ελεύθερο. Ε, χρειάζεται ποιοτικός ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά. Πέρα από το σχολείο ξέρουμε ότι εκεί εντοπίζονται πάρα πολλά προβλήματα. Τις διακοπές παραδείγματος χάρη Βλέπουμε παιδιά από εύπορες ε, οικογένειες ε, που έκαναν κάποια ενδιαφέροντα μαθήματα, έχουν περάσει πάρα πολύ ωραίε ε, διακοπές και μπορούν ευκολότερα να αφομοιώσουν αυτά που έμαθαν στο σχολείο πριν τις διακοπές. Το αντίθετο συμβαίνει με τα παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης πως υπάρχει και το φαινόμενο ε, αυτών που ε, το φαινόμενο της διάκρισης κατά αυτών που παίρνουν κοινωνικά επιδόματα θεωρούνται, θεωρείται ότι είναι υποδέστεροι. Σας ευχαριστώ. Κύριε Τουρ. Χαίρομαι που μπορώ να συμμετάσχω στην ενδιαφέρουσα και σημαντική συζήτηση. Είναι πολύ ε, σκοτεινές οι στατιστικές που δείχνουν πόσο μεγάλη είναι η παιδική φτώχεια και ο κοινωνικό αποκλεισμό. Στην ίδια μου τη χώρα 10% των παιδιών το 2012 ήταν σε απόλυτη φτώχεια. Παρόλο που ε, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο η χώρα μου θεωρείται ε, μια επιτυχής ιστορία. Πρέπει να θεσπιστεί το πλαίσιο για καλύτερη συνεργασία. Αλλά νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα εντείνει την πολιτική πίεση που ασκεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις χώρες μέλη για να αρχίσουν, να προχωρήσουν δηλαδή σε μια ουσιαστική συνεργασία για την καταπολέμηση παιδικής φτώχειας στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το πιο σημαντικό βήμα ίσως θα είναι να υιοθετηθούν ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές υπέρ των παιδιών σε όλες τις χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Γκέρκε. Όταν μιλούμε για παιδική φτώχεια εδώ, μιλούμε βεβαίω και για φτώχεια των γονιών. Χαίρομαι που ξεκαθαρίσατε το θέμα, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό, ειδικά εδώ, να τεθεί ως θέμα. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ μου είπε ότι υποστηρίζει μια ευρωπαϊκή οικογενειακή στρατηγική και νομίζω ότι κάτι μπορεί να βγει από αυτό. Όταν μιλούμε για παιδική αλλά και γονική φτώχεια, μιλούμε για κάτι το οποίο σημειώνεται και συνεχίζεται εδώ και πολλές γενναίες. Μιλούμε δηλαδή για αποτυχία της πολιτικής και όχι βεβαίως τα τελευταία 10 χρόνια, ίσως και τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα θεμελιώδες πρόβλημα μπροστά μας. Όταν μιλούμε για φτώχεια των γονιών ή ιδίως των παιδιών. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, αλλά να έχουμε και συνείδηση του γεγονότος ότι τα θέματα αυτά που πάμε να επεξεργαστούμε τώρα χρειάζονται τουλάχιστον μια δεκαετία για να δείξουν τις πρώτες επιτυχίες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας ημών των πολιτικών. Δεν έχουμε στη διάθεσή μας 10 χρόνια, το πολύ 4 ή 5. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα σε μια πολύ ευρύτερη φάση, όχι μόνο παιδεία, όχι μόνο οικογενειακή πολιτική. Εγώ θα έλεγα κανένας νόμος να μην ψηφίζεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χωρίς να ελέγχεται για το εάν ενδεχομένως οδηγεί σε κάποια δυσμενή επίπτωση σε βάρος παιδιών και γονιών. Και γιατί άραγε αυτό να μην ισχύσει και για τις χώρες μέλη. Κάτι τέτοιο νομίζω θα κάνει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο πολύ φιλικότερη απέναντι σε παιδιά και οικογένειες κλπ. Και δεν θα χρειάζεται να φοβούμεθα την παγκοσμιοποίηση. Γιατί θα έχουμε μια στέρεη βάση η οποία θα αποτρέψει τη φτώχεια και τις μελλοντικές γενναίες. Ευχαριστώ Στάιν Ρουκ. Πρώτα θερμές ευχαριστίες προς τις προσκεκλημένες μας. Επαναλάβατε πολλές γνωστές πληροφορίες, αλλά προσθέσατε και νέες. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι η καταπολέμηση της παιδικής στόχιας βεβαίως δεν σημαίνει... Εδώ μιλούμε για τους πόρους που χρειάζεται η Ευρώπη για το μέλλον της και αξίζει να εγκύψουμε πολύ εκτενέστερα στο θέμα. Ειδικά δε η υπόδειξη σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις όλων των νομοθετημάτων, ακόμη και των ψηφοφοριών που διεξάγουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Οι επιπτώσεις λοιπόν σε παιδιά και οικογένειες οφείλουν, οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη. Να ξεφύγουμε δηλαδή από τις συζητήσεις βιτρίνας όταν μιλούμε για φτώχεια. Να ξεκινήσουμε υπερκομματικά μια προσέγγιση και εμείς ως σοσιαλδημοκράτησες και σοσιαλδημοκράτες στην ακρόαση των επιτρόπων προωθήσαμε την ιδέα μιας εγγύησης υπέρ των παιδιών, όπως εκείνη η εγγύηση για τους νέους. Η ερώτηση προς τις προσκεκριμένες μας είναι ποια θα ήταν τα πιο κέρια στοιχεία που χρειάζεται μια τέτοια εγγύηση υπέρ των παιδιών. Βεβαίως μιλήσατε και για τη σημασία της παιδείας για την καταπολέμηση της φτώχειας. Υπάρχουν ολόκληρες ευρωπαϊκές περιφέρειες που προσφέρουν δωρεάν παιδεία από την αρχή, δηλαδή από τον βρεφικό ή παιδικό σταθμό μέχρι και το πανεπιστήμιο. Θεωρείται ότι αυτό μπορεί να είναι ένα κλειδί, δηλαδή η πρόσβαση σε δωρεάν παιδεία μπορεί να είναι ένα κέριο στοιχείο που να βοηθήσει στην καταπολέμηση της φτώχειας. Να ενθαρρύνουμε λοιπόν τις χώρες μέλη, έστω και αν η παιδεία δεν εμπίπτει στις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαρτάν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταγγέλουμε τη φτώχεια των παιδιών, αλλά όπως αναφέρθηκε διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για την συνέπεια της πολιτικής λιτότητα στην ευρωπαϊκή πολιτική εδώ και ε, δεκαετίες και γι' αυτό είναι πάρα πολύ ενισχυτικό. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον μας, το μέλλον των εθνών μας. Όμως θα πρέπει να απαντήσω στον εκπρόσωπο ε, της μη οργάνωση που έκανε πολιτική τρόπο που μίλαγε για λαϊκίστικα κινήματα και για κινήματα της άκρας δεξιάς. Συντόμως πρέπει να πούμε ότι η φτώχεια δεν εντύπωση ότι είναι κάτι το μοιραίο, κάτι το οποίο αφορά την κακή ανατροφή των παιδιών από πλευρά των γονιών. Ναι, αλλά να σα πω ότι είναι το δικό μου πατέρα, ο οποίο προερχόταν από Εβραιοπολωνέζικη οικογένεια, οι οποίοι έφυγαν από την ε, Πολωνία να ξεφύγουν στο τέλος του 19ου αιώνα το Πογκρόμ. Και ε, ε, αυτά γίνανε το, 19, δηλαδή μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ζούσαν στο, στο στο στάβλο μέσα πάνω σε χώμα κοιμόντουσαν και ζητωνόντουσαν από τις αγελάδες και τις κοπρίες οπότε είδατε πως μεγαλώσαμε το 45 επομένως τα πήγε καλύτερα και επομένως αυτό δεν τον εμπόδισε να αναθρέψει τα παιδιά του. Και να, που βρέθηκα εγώ σήμερα και σας απαντώ αυτή τη θέση. επομένω βλέπετε ότι η φτώχεια δεν είναι κάτι το μοιραίο και δεν προέρχεται αναγκαστικά από την ανατροφή των φτωχών γονιών. Πέραν αυτού, αγαπητέ, το θέμα είναι ότι εσείς λέτε για αρρωγή με κάποιο τρόπο, λέτε για αυτό την πολιτική του Γκισέ, για αυτούς που ωφελούνται σε εισαγωγικά ε, ναι, αυτό είναι η γνώμη σας, αλλά νομίζω ότι μέσω της εθνικής εκπαίδευσης σε κάθε ε, χώρα υπάρχει, υπάρχει δωρεάν παιδεία, οπότε εκεί μπορούμε να καταβάλουμε κάποιες προσπάθειες και μπορεί ο καθένας να βρει αυτό το οποίο του αξίζει δουλεύοντας. Οπότε, τι να σας πω, ε, είπατε λίγο απ' όλα, αλλά από την άλλη μεριά είπατε για παιδιά φτωχών γονέων, για παιδιά μεταναστών. Μπρο, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί έτσι μου δίνει την ευκαιρία να σας πω για μένα που είμαι λαϊκιστής, κύριε, ότι τα πρώτα θύματα των ε, μετα... μεταναστεύσεων είναι οι μετανάστες και τα παιδιά τους. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Schultz. Κύριος Σούλτς. Ευχαριστώ και εγώ για τη διοργάνωση της ακροάσεως σήμερα το απόγευμα, την οποία βρίσκω σημαντική και βρίσκω άλλωστε πολύ θετικό που συζητούμε διεξοδικά το θέμα αυτό. Ήδη κάποιοι ευρωβουλευτές συνέβαλαν με σημαντικές παρατηρήσεις. Είμαι και εγώ πατέρας δύο παιδιών. Επιτρέψτε μου να πω και εγώ δύο λόγια. Προέρχομαι από μια γερμανική περιφέρεια όπου κατά τη γνώμη μου γίνονται πολλά πράγματα στο οικονομικό επίπεδο υπέρ των παιδιών. Και είμαι πεπισμένος ότι τα λεφτά και μόνο δεν μπορεί να είναι ο σωστός δρόμος για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ακούμε σήμερα. Για μένα είναι επίσης πολύ σημαντικό, ανεξαρτήτως του αν βγάζουν πολλά λεφτά οι γονείς ή όχι, να γνωρίζουν οι γονείς ότι εφόσον αποκτήσουν παιδιά, αναλαμβάνουν μια ευθύνη και ότι οφείλουν να φροντίζουν τα παιδιά και στη Γερμανία, παριμήν, και στην περιφερειά μου, υπάρχουν γονείς η οικογένεια όπου το μόνο μέλος της οικογένειας που σηκώνεται νωρίς το πρωί από το κρεβάτι είναι το παιδί που θα πάει στο σχολείο. Εκεί δεν μπορεί να βοηθήσει το κράτος, έστω και αν δώσει χρήματα. Πρέπει η οικογένεια να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεύτερο, η κυρία Στάινρουκ ε, μίλησε σχετικά. Στην περιφέρεια μου, Σαξονία Ανχάλτ, μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά 10 ώρες την ημέρα δωρεάν στον παιδικό σταθμό όταν οι γονείς έχουν ε, χαμηλό εισόδημα ή είναι άνεργοι. Παρ' όλα αυτά, στην περιφέρειά μου διαπιστώνονται προβλήματα παιδικής φτώχειας, επίσης ανισότητες ευκαιριών. Έτσι λοιπόν και στην εντό εισαγωγικών πλούσια Γερμανία υπάρχουν προβλήματα. Αν και βεβαίω η παιδική φτώχεια ορίζεται διαφορετικά παροιμήν από τι άλλε χώρε. Άλλωστε, έχω και προσωπικά την εμπειρία ότι είμαι και τόσο ηλικιωμένο βέβαια. Το πιο σημαντικό για την παιδεία του παιδιού είναι να έχει πρόσβαση στην παιδεία. Ανεξαρτήτως αν προέρχεται από οικογένειε με υψηλό ή με χαμηλό εισόδημα. Ευχαριστώ. Κρασναντεύσκη. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν θα μιλήσω για την παιδική φτώχεια. Είναι σημαντικό το ζήτημα, όμως θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που είπε ο συνάδελφος για τα πογκρόμ στην Πολωνία, αν κατάλαβα καλά. Δεν υπήρχε Πολωνία το 19ο αιώνα, δεν ήταν ανεξάρτητη χώρα τότε. Μάλλον εννοούσατε τα πόγκρομ σε αυτό που είναι τώρα επικράτεια της Ουκρανίας ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είναι ρωσο-ουκρανικό το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας ε, να μην υπάρχουν ε, παρανοήσεις και συγχύσεις σε σχέση με ιστορικά δεδομένα. Ευχαριστώ. Κυρία Τσούμπερε, θέλετε να κάνετε κάποιες καταληκτικές ε, παρατηρήσεις. Έχετε λίγα λεπτά. Μπορούμε να υποβάλουμε ερωτήματα ακόμη στους ομιλητές του πάνελ, έτσι δεν είναι. Θα, θα, απαντήσουν, έτσι, θα τους δώσετε τη δυνατότητα να απαντήσουν. Δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Συγγνώμη, έχουμε πάνω από 20 λεπτά μέχρι τις 4.30. Σχεδόν 20 λεπτά από εμάς 4.30 είναι ο προβλεπόμενος χρόνος αλλά έχουμε άλλα προβλήματα. Έχουμε πάρα πολλά ε, θέματα στην ημερήσια διάταξη. Φυσικά, αν θέλετε να υποβάλλετε μία ερώτηση, ευχαριστώ και να σας δώσουν απάντηση για να κλείσει το θέμα. Η κυρία Τσούμπερ, εγώ συμφωνώ με κάτι που ανέφεραν ε, όλοι οι ομιλητές, η κατανομή του πλούτου. Αυτό που βιώνουμε και κανείς δεν μπορεί να είναι διάφορος είναι ότι ε, τη σήμερον ημέρα κάποιοι παρά την κατάσταση αυτή ε, πλουτίζουν. Εξακολουθούν να πλουτίζουν. Ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, πολιτικές ανυπόφορες, ε, χρειάζονται περικοπές σε όλους τους τομείς. Είναι αδύνατο για χώρες όπως η Πορτογαλία, παραδείγματος χάρη, να αντιμετωπίσουν τα τοκοχρεολύσια και ταυτόχρονα να έχουν μια κοινωνική πολιτική. Δεν μπορεί τα τοκοχρεωλήσια να είναι υψηλότερα από τρει δαπάνε του ε, τομέα της υγείας στην Πορτογαλία είναι θέμα κατανομής ε, του εθνικού πλούτου. Ε, μιλήσατε επίσης για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Θα ήθελα να σας πω και το έχω αναφέρει και στο παρελθόν πως δεν είναι δυνατόν να κάνουμε συστάσεις και αφενός να λέμε πρέπει να μειώσουμε, να καταπολεμήσουμε την παιδική φτώχεια και ταυτόχρονα ζητάτε να εφαρμοστούν κανόνες που είναι ακριβώς αυτοί που εμποδίζουν την υλοποίηση αυτών των στόχων. Χρειαζόμαστε κοινή λογική. Δεν γίνεται να κάνουμε κάτι και το αντίθετό του ταυτόχρονα. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Αυτό φυσικά θα το αναφέρω στην έκθεσή μου. Δύο ερωτήσεις ε, για τα επιδόματα για τα παιδιά, τα δελτία ή τις εγγυήσεις, όπως θέλετε πείτε, τις εγγυήσεις για τα παιδιά. Θέλετε ε, να είναι καθολική στήριξη, δηλαδή ανεξαρτήτως εισοδήματος των γονέων ε, προτείνεται μια ομοιόμορφη εγγύηση η οποία θα πηγαίνει στο παιδί το ίδιο. Και επίσης ε, ποιους ε, κοινωνικού δείκτες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να περιορίσουμε την παιδική φτώχεια πέρα από του δείκτες που χρησιμοποιούμε στη Eurostat. Ποιοι είναι εκείνοι οι δείκτες ε, που μπορούν να καλύψουν ευρύτερα το θέμα της παιδικής φτώχειας και μπορούν να καλύψουν άλλες μεταβλητές. Παραδείγματο χάρη το ευζήν του παιδιού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα έχει ο καθένας δύο λεπτά για να προσπαθήσει πάρα πολύ σύντομα να απαντήσει τις ερωτήσεις της κυρία Ζούμπερ ή τυχόν άλλες ερωτήσεις που θεωρείτε ότι είναι σημαντικές από πλευρά των βουλευτών. Κύριε Hainsworth, από την Eurogel έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό ότι πρόκειται για ένα θέμα που αποσχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζεται σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό από τα κράτη-μέλη το πώς θα, θα τους συμπεριφερθούμε των παιδιών, τι θα κάνουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό και αφορά τις αξίες και το μέλλον μας. Υπάρχει μεγάλη προβληματική για την φτώχεια ε, των ενηλίκων και των ανηλίκων. Γιατί ε, ε, κοιτάξτε μέσα από τα μάτια των παιδιών τη φτώχεια τους τότε θα δείτε τις οικογένειες, τις κοινότητες, τα σχολεία, την υγεία τους. μην το πάρουμε διασπαστικά, αλλά είναι σημαντικό να δούμε την ε, οπτική γωνία των παιδιών. Και σας παραπέμπω στην σύμβαση του ΟΗΕ. Αυτή θα πρέπει να μας καθοδηγεί. Έχουμε και τη σύσταση επομένω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να την υλοποιήσουμε τη σύσταση αυτή. Αν το είχαμε κάνει τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά για τα παιδιά μας σήμερα. Πρόεδρος. Κυρία Σεν από την UNICEF να δώσω τη σκητάλη στον Ντόμινικ Ρίτσαρτσον ή την Ντόμινικ Ρίτσαρτσον τέλο πάντων γιατί θέλω να πω ότι ο Προβάς UNICEF είναι πάρα σημαντικό να έχουμε δείκτες για τα στερημένα παιδιά. Στον αφορά δηλαδή το εισόδημα το 2009 το 2014. Οπότε παρακαλώ η Eurostat να εξωθεί στα κράτη-μέλη κάθε χρόνο να συλλέγουν τα σχετικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σμολένσκι από το Save the Children, Save the Children. σώστε τα παιδιά. Από και από δική μα πλευρά, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με του προλαλήσαντε και για μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υλοποιηθεί αυτή η σύσταση σε σχέση με τι επενδύσει για τα παιδιά. Πρώτα πρώτα προβλησιμότητα στου πόρου, ο πρώτο πυλώνα, το οποίο έχει να κάνει και με του γονεί και με τι οικογένειε και δεύτερον στο να υπάρχουν ποιοτικέ υπηρεσίε. Ε, εγκάρσιο και οριζόντια για όλες τις πολιτικές, δηλαδή υγεία και παιδεία και στέγαση. Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε στα παιδιά κάποιες δυνατότητες. Τους πιο ευάλωτους να υποστηρίξουμε, τους μη προνομιούχους, αλλά να μην στιγματίζονται. Άρα θέλουμε οριζόντιες λύσεις. Και όσον αφορά τους δείκτες τώρα, έχουμε κάποιες προτάσεις για το πώς θα παρακολουθήσουμε ε, κλείνει το μικρόφωνο την πλευρά την πολυδιάστατη τέλος πάντων να δούμε τι γίνεται με κάποιους δείκτες που δεν αφορούν γνωστικά γνωστικές δεξιότητες τις δεξιότητες μέσω της ποιότητας της κοινωνικής ζωής ε, των πολιτικών δραστηριοτήτων κλπ. ποιότητα για των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και τους δείκτες που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στις ποιοτικές υπηρεσίες και το αποτέλεσμα που φέρνει αυτό οπότε και αυτοί οι δείκτες είναι δυνατόν να επιλεγούν καλύτερα με την εμπλοκή των παιδιών σε αυτή τη διαδικασία από το δίκτυο κατά της στόχες. Θέλω να πω κάτι στη συνέχεια κάποιου βασικού θέματος που είπαμε, σχέση με την οικογένεια και την φτώχεια των ανηλίκων. Είναι πολύ βασικό το θέμα της ε, κατανομής, συστημική προσέγγιση. Για όλους να μειωθεί η φτώχεια. Να μην εστιαστούμε μόνο στους γονείς. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα των ανηλίκων. Γιατί μιλούμε τώρα για την ευημερία των ανηλίκων. Πώς θα εξασφαλίσουμε να υπάρχει αυτό. Εκεί θα πρέπει να στρατευτούμε. Άρα προσέγγιση προς την οικογένεια αλλά να μην είναι ε, αυτή η μόνη κατεύθυνση που θα πάρουμε. Άρα να δούμε και τα θέματα που πλευρά των παιδιών. Κατά δεύτερο λόγο, έχουμε το θέμα των εγγύσεων. Πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Αλλά προσοχή να μην βιαστούμε. Να μην κάνουμε μία λύση στο γόνατο. Να είναι ολοκληρωμένη η λύση. Και όπως είπαν και οι συνάδελφοι, έχουμε αυτή την τόσο ε, δόκιμη, τόσο πετυχημένη σύσταση που κάνει τόσα πράγματα, μισθούς, ε, κοινωνική πρόνοια, υπηρεσίες, στέγαση, όλα αυτά και άλλα. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν μια δέσμη και να μην θεωρήσουμε ότι ε, ένα μέσο θα λύσουμε ένα πρόβλημα. Σολεντάρ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούμε σχεδόν με όλα όσα ακούσαμε είναι κοινωνικό πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Χρειαζόμαστε δική στρατηγική, θα πρέπει το πρόβλημα να το εντάξουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο στρατηγική. Το ρίσκο είναι ότι αν δεν συνεχίσουμε με τη στρατηγική ενώ του 2020, εάν αρχίσουμε να έχουμε θεματολόγια χωριστά, τότε δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις, αποτελέσματα, θα είναι λάθος το μήνυμα και οι απαντήσεις σε αυτούς που αμφισβητούν το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ναι, έχουμε κάποιες ε, επιλογές που έχουν σχέση με τα θεσμικά όργανα, όμως θα πρέπει να υπάρχουν τα σωστά αποτελέσματα και αντιμετώπιση της, ε, του γενικού αποκλεισμού, ε, της οπαστικοποίησης και του λαϊκισμού. Θα πρέπει να έχουμε οριζόντιες εγκάρσεις λύσεις για όλες τις χώρες, να επενδύσουμε στην παιδεία όπως ελέγχθη να έχουμε τις ε, υπηρεσίες σχετικές με παιδεία και κοινωνική πρόνοια. Έχουμε 150.000 κάποιο δίκτυο που ανήκει σε εμάς, ε, οι οποίοι είναι όλοι εθελοντές. Άρα, να μην θεωρείτε ότι όλα αυτά έχουν κάποια στροβουλία. Είναι στράτευση, ε, δέσμευση στα γαλλικά. Οπότε, νέο ναι, όπως είπατε, είναι θέμα δουλειάς, είναι θέμα παιδείας. Ναι, όντως όταν κάποιος κάνει το καθήκον τον μπορεί να ε, επικρίνει. Και αυτό ισχύει όμως και όταν κάποιος ε, δουλεύει μέσα σε, σε κάποια οργάνωση που κάνει τη δουλειά της και που λέγεται Solidar και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ευχαριστούμε και ο κύριος Ρίτσαρσον τώρα από τη UNICEF. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ε, η παιδική φτώχεια δεν είναι κάτι καινούριο, είναι διαγενειακό πρόβλημα. 30 ε, χρόνια ε, παρατηρείται το φαινόμενο, ταυτόχρονα με τις μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν τελεσφορήσει. Όμως κατά κάποιο τρόπο πρέπει να υπερπηδήσουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι δύο διαφορετικά διακριτά ζητήματα, γονεακή φτώχεια και παιδική φτώχεια. Όντω έχουν την ευθύνη τα οι γονείς, αλλά δεν επιλέγουν τους γονείς τους τα παιδιά ε, και η κοινότητα και η κοινωνία πρέπει να φροντίζει τα παιδιά. Το ζήτημα της πολιτικής είναι περίπλοκο. Οι, πιο, οι χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη επιτυχία έχουν ε, χαμηλά επιδόματα αλλά καθολικής πρόσβαση. Επίσης έχουν καθολικά αλλά όχι δωρεάν ζητήματα, περί, ε, συστήματα συγγνώμη, περίθαλψης των παιδιών, φύλαξης των παιδιών ε, και... Ευχαριστώ πηγαίνουν κάποιοι στην αγορά εργασίας, ε, με, ε, κάποιοι που έχουν υψηλά εισοδήματα, παρόλα αυτά έχουν δωρεάν περίθαλψη και καταλαβαίνετε ότι είναι αντίστροφα τα αποτελέσματα από τα επιθυμητά. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε όταν ε, θέλουμε να συμμετέχουν περισσότερο οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, να προστατεύσουμε τα παιδιά, να είμαστε προσεκτικότεροι με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε. Ε, οι καλύτεροι δεν είναι αυτοί που έχουν τις υψηλότερες δαπάνες. Ε, θα ήθελα να το προσέξουμε αυτό επίσης. Στην Ευρώπη, τρία από κάθε πέντε ευρώ τα δαπανούνται για τα σχολεία, αλλά όχι για την ηλικία μέχρι, τα, ε, μέχρι έξι χρονών. <coughs> Τι γίνεται λοιπόν στην αρχή της ζωής ε, του παιδιού. Θα πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά, διότι εάν δεν έχουμε προετοιμάσει τα παιδιά για το σχολείο και τα σχολεία για τα παιδιά, τότε ε, δεν βελτιστοποιείται η επένδυση που γίνεται. Και γι' αυτό νομίζω ότι χρειαζόμαστε νέους διεκτές ούτως ώστε να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της διαγενειακής έλλειψης κινητικότητας, ανισότητας και φτώχειας. Θα πρέπει μέσα στο σχολείο να στηρίξουμε τα παιδιά για να αξιοποιήσουν πλήρως αυτή τη δυνατότητα, να ολοκληρώσουμε τις υπηρεσίες υγείας στα σχολεία ούτως ώστε να υπάρχει υποστήριξη για τα παιδιά στη μειονεκτικότερη θέση και ένας δείκτης ε, για τα άπορα παιδιά που θα χρησιμοποιείται για την χορήγηση υπηρεσίας υπηρεσιών στα παιδιά. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα ολιστικό μέτρο, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Σας ευχαριστούμε για τις ε, ε, απαντήσεις σας. Σίγουρα θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια αυτό το ζήτημα. Κλείνει η συζήτηση για αυτό το σημείο και περνάμε στο σημείο 10 ε, της Μέσης Διαταξής «Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη». Πρόκειται για ένα σχέδιο χνομοδότησης. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Πρεσναντεύσκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται όντως για γνωμοδότηση. Αυτό αντιλαμβάνεστε μας περιορίζει, διότι είναι περιορισμένος ο χώρος σε σελίδες που δίνει ο κανονισμός του Κοινοβουλίου. Πρώτα όμως θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και εισηγήτριες για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που μου έχουν υποβάλει. Βέβαια δεν χωράνε όλες σε αυτό το σύντομο κείμενο. Ως πανεπιστημιακός έχω συνηθίσει άλλωστε να συγγράφω πολύ μακροσκελέστερα κείμενα και γνωμοδοτήσεις, αντιλαμβάνεστε. Τι θα βάλω τώρα στη γνωμοδότηση. Πρώτα, τη σημασία βέβαια των οικογενειακών επιχειρήσεων. Επίσης από τις διάφορες μελέτες περιπτώσεων και στάντης των οικογενειακών επιχειρήσεων αντλούμε κάποια συμπεράσματα. Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν ένα σύστημα αξιών που υπαγορεύει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν καθημερινά, σε καθημερινή βάση. Νομίζω ότι από αυτού σημειώνεται συνένεση, διότι σε όλους μας αρέσουν αυτές οι αξίες, όπως για παράδειγμα η δέσμευση υπέρ των τοπικών κοινωνιών. Η παράδοση αυτή του ε, έντιμου εμπόρου. Ε, παρακάτω, επισημαίνω το γεγονό επίσης ότι ο ίδιος ο ορισμός της οικογενειακή επιχείρησης στερείται σαφήνειας. Δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρο ορισμός. Πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη και τις διαφορές μεταξύ των χωρών μελών. Θα πρέπει ωστόσο να, να καταθέσουμε ένα σχέδιο ορισμού τουλάχιστον. Γιατί τότε θα είναι ευκολότερο και για μα, τουλάχιστον να μπορέσουμε να συλλέξουμε πληροφορίε σχετικά με αυτό το είδο επιχειρήσεων. Σημαντικό είναι επίσης να τονιστεί η ανάγκη εκπαίδευσης, γιατί συχνά οι οικογενειακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον τρόπο που διαχειρίζονται την κληρονομιά της επιχείρησης. Συχνά άλλωστε οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Και βέβαια η οικονομική κρίση και η ύφεση οδήγησαν σε δύσκολους καιρούς για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Και αυτό που εμείς θα θέλαμε να δούμε είναι ανάληψη δράσης από τον πρόεδρο Γιούνκερ δεν μπορεί να λησμονήσει τις οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι σημαντικός στήλος της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας σε όλες τις χώρες μέλη και πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό. Τέλος δε. Περιλαμβάνουμε και περιλαμβάνω δηλαδή σχόλια σχετικά με τα όσα έχω μάθει για τις διαρροές του Λουξεμβούργου, τα Lux Leaks. Χρειάζεται ισότιμη μεταχείριση πολυεθνικών και μικρών επιχειρήσεων, οικογενειακών επιχειρήσεων κλπ. Σε αυτό αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην τελευταία παράγραφο της γνωμοδότησης. Βεβαίω υπάρχουν χώρες όπου μετά το 1945 εξαφανίστηκαν στην ουσία οικογενειακές επιχειρήσεις. Αλώθηκε η οικογενειακή επιχείρηση εξαφανίστηκε, καταστράφηκε. Αυτό συνέβαινε από την μια μεριά. Από την άλλη μεριά, σε άλλες χώρες, εποφελήθηκαν οι οικογενειακές επιχειρήσεις από αλλοδαπές επενδύσεις. Και προχώρησαν, μεγάλωσαν. ακόμα και με τη συνθήκη της Βασοβίας προβλεπόταν στήριξη για τις επιχειρήσεις. Πάντως δεν έχουμε δει κατάσταση όπου οι οικογενειακές επιχειρήσεις να είχαν ενισχυθεί. Αντιμετωπίζουν βέβαια και προβλήματα με τη φορολογία, γιατί αντίθετα με τις με τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους που μπορούν και φόρο αποφεύγουν, οι οικογενειακές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή. Θα συντάξουμε και τροπολογίες και αναμένω βέβαια και τις συζητήσεις που θα διεξαγάγω με τους και συζητητές και με τους υπολείπους συναδέλφους. Κύριε Κοσλόφσκα εκπροσωπείτε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εσείς στη θέση του ή της ε, σκιώδους εισηγήτριας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει κυρία Κοσλόφσκα. Κυρία Γιασλοφσιέσκα, όντως είναι η σκιώδη προεδρε λεει κυρια κοσλοφσκα κυρια η αλλά δεν μπόρεσε να παραστεί και θα μιλήσω για λογαριασμό της και εκ μέρους της. Οπότε, συγχαρητήρια γιατί είναι πάρα πολύ καλή αυτή η έκθεση. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την οργάνωση αυτήν την ε, συνάντηση και ευχαριστούμε για τον τρόπο που εργάστηκε. Οπότε ε, είμαι βέβαιος ότι όλοι θα συνεχίσουν την ε, επικοδομική συνεργασία. Μια που οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, είναι μια παράδοση, είναι κάτι που να συνεχίσουμε, το στηρίζουμε. Βέβαια είναι και θέμα ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ομάδας εμπειρογνωμόνων πρότεινε να υπάρξουν κάποιες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το εμπορικό δίκαιο αλλά και το φορολογικό δίκαιο για να βοηθηθούν ακριβώς οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Πολύ σημαντικό και επίσης όσον αφορά ε, αυτά τα στοιχεία τα, εκπαιδευτικά. Το 2009 είχαμε κάποια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα με αυτήν σε πολλά κράτη-μέλη είχαμε αυτοπασχολούμενους οι οποίοι ίδρυαν κάποιες εταιρείε. Αυτές θεωρούνται οικογενειακές επιχειρήσεις και ήταν πάρα πολύ σημαντική η επίδρασή τους στις οικογένειες. Υπήρχε και θέμα μετά ε, στο κληρονομικό δίκαιο, υπήρχε θέμα μεταβίβασης στις επόμενες γενναίες των στοιχείων του ενεργητικού αυτής της περιουσίας, Οπότε αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει είναι να έχουμε μια σωστή ρύθμιση και εγώ θα κατεβάσω και μια σχετική τροπολογία σχετικά. Ο κύριος ε, Μπενίφη για το σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο κειμένου για τις γενικές επιχείρησεις. Απ' την αρχή φάνηκε ότι έχει πνεύμα συνεργασίας για όλους τους εισηγητές. Είναι καλή ευκαιρία αυτή. Να συμβάλλουμε σε αυτό το έγγραφο να είναι ενημερωμένο, να καλύπτει αυτόν τον κλάδο που συμβάλλει πάρα πολύ στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Πάντως θα πρέπει να σταθούμε στο ότι δημιουργούνται θέσεις απασχόληση από αυτές τις επιχείρησεις στις, ε, στην καλή παράδοση που υπάρχει, ε, στη βιωσιμότητα που έχει δείξει ότι έχει, που πάει καλύτερα αυτός ο κλάδος από ό,τι άλλοι κλάδοι της οικονομίας και επίσης που είναι προσανατολισμένος αυτός ο κλάδος σε μακρόπνοη ανάπτυξη. Επομένως, το κείμενο αυτό είναι μια καλή αρχή. Και πρέπει επομένως με αυτό το πνεύμα να δουλέψουμε. Τώρα, κάποιες άλλες παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να καλυφθούν. Μακάρι να εμπνεύσουν και τη δουλειά μέσα εδώ. Σωστά, ο εισηγητής θέτει το ζήτημα του ορισμού τις επιχείρησεις αυτές. Αφού όμως έχουμε δεδομένο το έργο της ομάδας Εμπειρονομών και του ευρωπαϊκού ορισμού από το 2009, γιατί τον δεδομένο αυτόν ορισμό να τον αλλάξουμε. Έχουμε κάποια κριτήρια, τα οποία κριτήρια δεν είναι στεγανά το τι είναι τέτοια επιχείρηση. Είναι θέμα κυριότητας της εταιρείας, είναι θέμα του ποιος αποφασίζει αν έχει άμεση με τις αποφάσεις, η έμεση, η, το μέγεθος της εταιρεία. Έχουμε διάφορες παραμέτρους, σύμφωνα τις οποίες θα μπορούσε κάποιος στην κεντρική Ιταλία να φτιάχνει ε, λουκάνικα, αλλά είναι κοινωνική επιχείρηση και το IKEA. Μα είναι και η Volkswagen. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να χτενίσουμε κάπως αυτόν τον ορισμό. Χρειάζεται να το κάνουμε αυτό εμείς ως νομοθέτες, αλλά και ο κλάδος το θέλει για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα τις ενεργειές μας και να έχουμε πιο δόκιμο νομοθετήματα. Οι επιχειρήσεις αυτές ε, δουλεύουν καλύτερα όταν έχουν κοινωνική υπευθυνότητα, όταν ωφελούν του ε, εργαζομένους αλλά και τι κοινότητε που είναι εγκατεστημένε. Αυτά τα αναγνωρίζει το σχέδιο κειμένου των συναδέλφων τη Επιτροπή Ήτρε που είναι πολύ θετική. Άρα θα πρέπει, μπορούμε αυτό να το πούμε όσον αφορά επομένω τα στάνταρ τη κοινωνική ευθύνη επίσης τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων στην κοινωνική επιχείρηση. Φαντάζομαι ότι θα, θα τα βρούμε, δεν θα διαφωνήσουμε. Τέλος, υπάρχει ένα στοιχείο γεωγραφικό που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη. Λέει ότι η κατανομή είναι άνηση αυτών των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχουμε διαφορετικές συνθήκες οικονομικές στην Ευρώπη. Θα πρέπει να μας προβληματίσει και αυτό το στοιχείο της γεωγραφικής κατανομής. Σας ευχαριστούμε κύριε Μονιφάη. Η Ρενάτε Βέμπερ τώρα Φιλελεύθερου. φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αληθεύει ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες για τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας για το μήκος, τους, το μήκος του σχεδίου έκθεσης και της νομοδότησης που εκδίδουν οι συναρμόδιες επιτροπές. Ταυτόχρονα όμως είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή διότι μια τέτοια έκθεση πρωτοβουλία ε, με τη συμβολή της Επιτροπής Αποσχόληση ε, συνιστά μια κοινή προσπάθεια εκπόνησης ε, κοινών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες θα οδηγήσουν σε καλύτερη νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα. Δεν αμφιβάλλω ότι στο πέρας αυτής της ε, περίπλογης διαδικασίας με τις ε, συσκέψεις και τις τροπολογίες θα έχει αλλάξει στο μεταξύ το σχέδιο γνωμοδότησης καθώς και η έκθεση ίδια. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το σχέδιο που συνέταξε δείχνει ανοιχτό πνεύμα στη συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές ως προς τις προτάσεις που θέλουμε να κάνουμε. Κατά πάσα πιθανότητα το σημαντικότερο ζήτημα είναι ο ορισμός της οικογενειακής επιχείρησης. Μια... Φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικά σενάρια και εγώ θα ήθελα στην, σε μια τροπολογία μου να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κοινού δείκτες που είναι απαραίτητοι για να ταξινομηθεί ως οικογενειακή μια επιχείρηση και ίσως τότε να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερα στατιστικά στοιχεία και μια σφαιρικότερη εικόνα για το ρόλο που διαδραματίζουν στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οικογενειακές επιχειρήσεις ε, ε, αλλά και το ρόλο τους στη, ως προς την απασχόληση. Η πολιτική ομάδα των φιλελευθέρων επιθυμεί να ε, ληφθεί υπόψη και το θέμα της ισότητας των δύο φύλων σε αυτό το τομέα. Θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες. Επίσης μας ενδιαφέρει η ιδέα της μονοπευθυντικής θηρίδας για τις γυναίκες επιχειρηματίες συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης για ε, τη φύλαξη των παιδιών για όσες γυναίκες θέλουν να δραστηριοποιηθούν ως επιχειρηματίες σε μια οικογενειακή επιχείρηση. Τι σημαίνει η μεταβίβαση της ηγεσία και η διαδοχή ε, στον τομέα των οικογενειακών επιχειρήσεων να είναι ένα σημαντικό σημείο. Εξίσου σημαντικό επίσης είναι το ότι αν θέλουμε να εξακολουθήσουν αυτές οι οικογενειακές επιχειρήσεις να διαδραματίζουν ένα δυναμικότερο, ένα πιο δραστήριο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, είναι σημαντικό να δούμε με ποιο τρόπο θα νομοθετήσουμε. θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να ενοποιήσουν και να απλουστεύσουν τα νομοθετήματα που ε, είναι σε ισχύ σε αυτό το τομέα. Ταυτόχρονα, εάν θέλουμε οι επιχειρηματίες των οικογενειακών επιχειρήσεων να είναι πιο δραστήριοι, θα πρέπει να ε, δράσουμε σε προγενέστερο στάδιο, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκεί θα αποκτήσουν προσόντα για να μπορέσουν να αναλάβουν ένα τέτοιο ενεργό ρόλο. Κλείνοντας, είμαι πεπισμένη ότι θα είναι πολύ καλή αυτή η γνωμοδότηση που σε συνδυασμό με την έκθεση θα μας βοηθήσει στην εκπόνηση της πολιτικής που χρειαζόμαστε. Κύριος Ηλικιώτης. Ε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την καλή δουλειά που έχει κάνει για σύνταξη αυτή της νομοδότησης. Οι θέσεις του εισηγητή του κύριου Κρασνοντεύσκη γίνονται πολύ ξεκάθαρες μέσα από το σχέδιο γνωμοδότησης κάνοντας έτσι δυνατή τη σαφή τοποθέτηση της κάθε ομάδας. Ως ΚΟΕ βεβαίως έχουμε σημαντικές διαφωνίες με τη γνωμοδότηση, με το σχέδιο γνωμοδότησης με κυριότερη αυτήν την εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικότητας στη σχολική εκπαίδευση. Η δική μας αντίληψη ως ομάδα είναι πως η εκπαίδευση πρέπει να απεμπλακεί από την οικονομία της αγοράς μέσα από τη διαμόρφωση ενός σχολείου ως δημοκρατικού σχολείου του πολίτη στο οποίο οι μαθητές, τα παιδιά δηλαδή και οι νέοι θα βιώνουν την παιδική και νεανική τους ηλικία ως τις πιο δημιουργικές και ευτυχισμένες περιόδους της ανθρώπινης ζωής η επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα ή ο οικονομικός δαρβινισμός δεν μπορούν να έχουν θέση εκεί, να έχουν θέση δηλαδή στο σχολείο. Άλλο σημείο το οποίο θεωρούμε πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης είναι στον ορισμό των οικογενειακών επιχειρήσεων. Συμφωνώ και με την σκιώδη εισηγήτρια από, από την Άρτην ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στα κράτη-μέλη ε, εμείς είμαστε της άποψη πω οι οικογενειακές επιχειρήσει πρέπει να διαχωριστούν, να διαχωρίζονται όπω ε, όλες οι άλλες επιχειρήσεις στι πολύ μικρές, τι μικρές, τι μεσαίε και τι μεγάλες ενώ θεωρούμε πρέπει να δημιουργηθεί μια κατηγορία για επιχειρήσεις μέχρι πέντε απασχολούμενους αφού τέτοιε επιχειρήσεις είναι στη συντηρητική του πλειοψηφία οικογενειακές επιχειρήσεις. Και σε αυτές τις επιχειρήσεις πρέπει να δίνεται βοήθεια στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση αλλά και άλλα κινητρά όπως για παράδειγμα μια δίκαιη προοδευτική φορολόγηση και διασφάλιση ρήτρων προστασίας τους. Πέραν όμω των διαφωνιών μα, χαιρετίζουμε τη δέσμευση του συγητή για σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων στι οικογενειακέ επιχειρήσει και κατανοούμε την ανάγκη για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω τη οικονομική κρίση. Αντιλαμβανόμαστε κι εμεί πω με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διασφαλιστούν θέσει εργασία. Ε, με προοπτική να δημιουργηθούν και καινούργιε. Είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των νέων θέσεων εργασία ε, δημιουργούνται από μικρομεσαίε επιχειρήσει, ε, που εκεί εντάσσονται και οι οικογενειακέ επιχειρήσει. με αυτέ τι σκέψει θα καταθέσουμε τι τροπολογίε μα και είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε ε, με τον εισηγητή σε παραγωγικό και επικοδομητικό πνεύμα ε, για βελτίωση της νομοδότησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you. Ε, Σας ευχαριστούμε. Η Τατιάνα Στανόκα από τους Πράσινους θα πάρει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Ναι, και για την ε, συνεργασία που είχαμε και αυτή την πρώτη συζήτηση πριν τις γιορτές ε, καταθέσαμε τις τροπολογίες μας. Θα ε, συζητήσω συντομία, μάλλον θα παρουσιάσω συντομία το περιεχόμενό τους και θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα στον εισηγητή στην παρουσίαση που κάνατε είδαμε κάποια διαφορετικά σημεία για τις πολυεθνικές παραδείγματος χάρη και για τις μικρές επιχειρήσεις. Ε, μιλήσατε για γεωγραφικό περιορισμό. Λέει μέσα το κείμενό σας ότι ζητάμε, ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίση μεταχείριση για τις οικογενειακές και για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Εμεί διαφωνούμε. Και εμείς λέμε τα εξή στην τροπολογία μας. Ευχαριστούμε την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι χρειάζεται στο ότι ε, ε, λοχεύει ένας κίνδυνος ε, αν υπάρξει ισότιμη μεταχείριση ανάμεσα στι οικογενειακές και πολυεθνικές επιχειρήσεις σε σχέση με την φοροαποφυγή λόγω της διαφοράς των πολυεθνικών με τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι περιορισμένες γεωγραφικά ως προς τη δράση τους. Κάνουμε και προτάσεις συμβιβασμού δεν νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε τόσο αισιόδοξοι δε, για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν ισχύει ότι είναι πάντοτε επιτυχημένες ε, στην αιτιολογική σκέψη ε, και εδώ έχουμε καταθέσει η τροπολογία. Λέμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ε, είναι επιτυχημένες οι οικογενειακές επιχειρήσεις και έχουν αυτή τη διαχρονική ε, στρατηγική και μακροπρόθεσμη επιτυχία. Για τον ορισμό των οικογενειακών επιχειρήσεων περιμένουμε ακόμη, δεν υπάρχει και όπως και η Ρενάτε από τους ε, φιλελεύθερους θα θέλαμε και εμείς να έχουμε κριτήρια ταξινόμησης των επιχειρήσεων ε, ως οικογενειακών. Έχουμε καταθέσει και μια άλλη τροπολογία όπου ζητάμε από την Επιτροπή όταν επεξεργαστεί τον ορισμό να λάβει υπόψη και την ποικιλομορφία των οικογενειών. Ε, στην ευρωπαϊκή κοινωνία και να μην υπάρχει καμία διάκριση κάποιων μορφών οικογένειας. Ε, έχουμε καταθέσει τροπολογία για την παράγραφο 2, ε, εκεί που μιλάτε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. εξηγούμε επακριβέστερα εδώ το πλαίσιο που είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στη δικαιοσύνη, κοινωνική προστασία όλων όσων εμπλέκονται σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. αναδιάρθρωση του τομέα της υγείας με επιπτώσεις στην ε, διατήρηση της θέσης εργασίας. Ε, αναφερόμαστε και στην κυκλική οικονομία πάλι σε σχέση με την διατήρηση ε, θέσεων εργασίας καθώς και ε, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Απλώς διευκρινίζουμε δηλαδή το περιεχόμενο αυτής της παραγράφου. Αναγνωρίζουμε βεβαίως ότι ε, είστε περιορισμένος ως προς το μήκος της νομοδότησης. Εμείς πάντως θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να είμαστε σαφέστεροι. Σας ευχαριστούμε και ο κύριος Γκερί και τώρα ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και πρώτα ευχαριστώ τον συνάδελφό μου καθηγητή Κραζονεύσκη για την θαυμάσια πρόταση ε, γνωμοδότηση που έχει φτιάξει αλλά και τη συνεργασία μέχρι εδώ. Για μένα στην γνωμοδότηση υπάρχουν δύο πράγματα που είναι σημαντικά. Η ευρωπαϊκή διάσταση του παραδοσιακού ορισμού του έντιμου εμπόρου. Honorable Merchant στα αγγλικά. Βρίσκω ότι το είδος αυτό είναι και, πώς να πω, απηχεί την παραδοσιακή ιστορία της οικογενειακής επιχείρησης. Και να μην λησμονούμε ότι αυτό πρέπει να προβληθεί και στην παγκόσμια αγορά. Ο έντιμος έμπορος θα πρέπει να γίνει το σήμα κατά τεθέν της Ευρώπης. Εκεί οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Από την άλλη μεριά, Το ζήτημα της φορολόγησης της κληρονομιάς, του φόρου κληρονομιάς δηλαδή, δεν είναι βεβαίω ευρωπαϊκό θέμα. Είναι σημαντικό όμως να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες μεταφοράς της περιουσίας από γενιά σε γενιά. Εδώ ο ευρύ συνασπισμός που ασκεί την κυβέρνηση στη Γερμανία θα πρέπει να ελαφρώσει το ε, φορολογικό βάρος στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Τελειώσατε, δεν είναι κύριε Κύριε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μορβάη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που στην έκθεση του ο συνάδελφός μου αναφέρεται και στις πρώην κομμουνιστικές χώρες και την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εκεί. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης είχε ιδιαίτερη σημασία στα κομμουνιστικά καθεστώτα το ανυπαρκτό σοσιαλισμό, όπως θέλετε πέστε το, η δημιουργία απασχόλησης γινόταν μόνο από τις μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις, μεγάλα εργοστάσια κρατικής ιδιοκτησίας. Μετά από την μετάβαση ήρθε κάτι το παρόμοιο, γιατί οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις δημιουργούσαν τις δουλειές. Ήρθαν στην Ουγγαρία, έφτιαξαν αλυσίδες παραγωγής και δημιούργησαν απασχόληση. Αυτή είναι η συνήθις, η οπτική. Θα πρέπει να αλλάξει όμως η οπτική αυτή. Οι κυβερνήσεις πρέπει να κατανοήσουν ότι και το ζευγάρι εκείνο που φτιάχνει μια μικρή οικολογική φάρμα, ένα αγρόκτημα και ζει εκεί με τα τρία παιδιά του και έχουν και ένα εργαστήρι και φτιάχνουν τυρί κτλ. Και, και φτιάχνουν έτσι μια μικρή επιχείρηση. Χρειάζονται και αυτή η υποστήριξη. Όχι μόνο να υποστηρίζουν τι μεγάλε πολυεθνικέ επιχειρήσει, με φορολογικές ελαφρύνσεις, με κρατικές επιδοτήσεις κτλ. Και αυτές οι μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν απασχόληση, απασχόληση αξιοπρεπή. Πρέπει να δημιουργηθεί με τον τρόπο αυτό μια μεσαία τάξη. Τότε θα μειωθεί η διαφθορά, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βεβαίως δεν θα εξαρτώνται από το κράτος και από τις πολυεθνικές και θα μπορούν να ελέγχουν το κράτο Μάλιστα. Ένα λεπτό ακόμα, ο ίδιο ο εισηγητή, κ. Κρασνογεύσκη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Μιλώντας για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, να μην ξεχνούμε τι είχε γράψει ο Τόμας και ο Μαξ Βέμπερ ότι ότι έχουμε πολλές οικογένειες, τέτοιες, συγγνώμη, επιχειρήσεις και εδώ και πολλά, πολλά χρόνια. Και φυσικά η επόμενη γενιά πρόκειται να κληρονομήσει την επιχείρηση. Επίσης, έχουμε αυτή τη στιγμή έναν υπερβολικά ευρύ ορισμό της οικογενειακής επιχείρησης. Ας πούμε, ο όμιλος επιχείρησεων Volkswagen αποτελεί οικογενειακή επιχείρηση. Από την άλλη μεριά. όλες οι κοινωνικές επιχειρήσεις θέλουν να είναι πετυχημένες, θέλουν να επεκτείνονται και αυτό να γίνεται από γενιά σε γενιά, να περνάει από τη μία γενιά στην άλλη αυτή η επιτυχία. Δηλαδή είναι προβληματικός ορισμός, πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Βεβαίω είναι και θέμα παιδείας και εκπαίδευσης και με εκπλήσουν αυτά που είπε ο συνάδελφος από την ΚΟΕ. Εγώ είμαι υπέρ της ε, παιδείας, αλλά αυτό σημαίνει και εκπαίδευση στο επιχειρηματικό πνεύμα. Δηλαδή κάποιο να είναι εφευρετικό, κάποιο που θέλει τελικά να γίνει επιχειρηματίας. Γιατί θυμάμαι πώς ήταν τα πράγματα στην Πολωνία όταν ήμουν μικρός. Είχαμε κάποιου εργαζόμενους που προσπάθησαν να στήσουν μια επιχείρηση όταν επιτράπηκε αυτό και προσπάθησαν να περάσουν γενικό πνεύμα εκεί. Μα ακριβώ και μπορεί να βοηθηθεί μια τέτοια επιχείρηση από την παιδεία. Τώρα, όσον αφορά τις ανισότητες, όπως ε, ακούσαμε από τους πράσινους, αυτές οι μικρές κοινωνικές επιχειρήσεις όντως δεν απολαύουν ισότητας. Βέβαια στη Γερμανία τα πράγματα ίσως είναι καλύτερα από ό,τι αλλού. Αλλά υπάρχουν διαφορές μεγάλες από χώρα σε χώρα. Λάβετε μόνος υπόψη αυτές τις διαφορές. Γιατί γίνεται δηλαδή στις χώρες της περιφέρειας της Ένωσης. Δεν υπάρχει καν κουλτούρα οικογενειακής επιχείρησης σε πολλές χώρες και αυτό τώρα πρέπει να το αλλάξουμε. Πάντως, όλα όσα είπατε νομίζω ότι είναι δημιουργικές ε, συμβολές στη συζήτησή μας και άλλωστε και εγώ πανεπιστημιακό ήμουν, έχω συνηθίσει διαφορετικές απόψεις, οπότε θα προσπαθήσω όσο μπορώ καλύτερα να σας καλύψω όλους το κείμενο. Thank you, Mr. The deadline for amendment... Η προθεσμία είναι η 14η Απριλίου, το μεσημέρι. Καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες. Μπορείτε να ενημερωθείτε και να ενημερώσετε από email σε σχέση με κάποιο αναφερμένο κείμενο. Και επίσης όλες και όλες τις άλλες πληροφορίες για τις τροπολογίες επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε. 7 Μαΐου πρόκειται να ψηφίσουμε το κείμενο. Σήμερα τώρα 11 σήμερα στη διάταξη έκθεση ή εκθέσεις όσον αφορά την αναλογικότητα και επικορικότητα για 2012 και 2013 πρώτη συζήτηση της ε, έκθεσης. Η κυρία Χέλγα Στίβενς είναι συγγύτρια και του δίνω το λόγο. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ. Είμαι η συγγήτρια για αυτό το ζήτημα. Είναι ένα σχέδιο έκθεσης μόνο. Ε, που θα υποβάλουμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, που τη Επιτροπής Απασχόλησης. Έχουμε ένα σχέδιο συστάσεων για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Θα ήθελα να κάνω μια επισκόπηση των συστάσεων. Η αναλογικότητα και η επικουρικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για την ομάδα μου. Καλωσορίζουμε την συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβουλία. Τονίζουμε ιδιαίτερα στη σημασία των τοπικών κοινοβουλίων, κυρίως δε αυτών που έχουν και νομοθετική εξουσία. Απευθύνουμε λοιπόν μια έκκληση για, ε, ε, ε, για ενεργότερη συμμετοχή τους στο σύστημα έγκυρης προειδοποίησης. Το Πολωνικό Κοινοβούλιο είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα Ε, διάφορα τοπικά κοινοβούλια στην Πολωνία έχουν υποδειγματική δράση. Η εξάντε αξιολογήσεις αντικτύπου πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να καταφθάνουν νωρίτερα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ε, συμπεριλαμβάνουμε αυτά τα στοιχεία στις νομοδοτήσεις μας είναι σημαντικό δε να ε, εφαρμόζουμε την αρχή του Think Small First ε, ούτως ώστε να μειώνεται και το κόστος για τις επιχειρήσεις και να προσθέτει η εφαρμογή της νομοθεσίας. Αυτή είναι η περίληψη των συστάσεών μας και θα ήθελα να ακούσω τώρα τις απόψεις και τις προτάσεις τις οποίες θα προσπαθήσω να ε, συμπεριλάβω. Μετά τις ε, διακοπές ε, θα οργανώσουμε και μια συνάντηση με τους σκιώδες εισηγητές. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοσλόσκα Ράντγεβης τώρα, η σχέση εισηγητρία από πλευράς του ΕΛΚ θα πάρει το λόγο. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και δεν μεταφράζεται η ομιλήτρια. Πρόκειται για το θέμα τώρα της αναλογικότητας. Οπότε, κατά τη γνωμοδότηση ζητείτε κάποιο είδους αναθεώρηση του κανισμού. Θέλετε να επαναλάβω. Ναι, γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα και δεν μεταφραζόταν, λέει, η πρώτη χωρίς μικρόφωνο. E, doceniając dotychczasową e, Θέλω να σας πω πάλι ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για το, έργο το οποίο έχει γίνει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά να καλύψουν και την αναλογικότητα και την επικουρικότητα που είναι πολύ σημαντικά. Όμως αυτό που επίσης χρειάζεται είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε το έργο της Κομισιόν που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει έναν ε, πολιτικό διάλογο. Παράλληλα με τον έλεγχο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτό επομένως μπορεί να είναι ένα μέσον πάρα πολύ χρήσιμο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αναλογικότητα και επικορικότητα. Ο πολιτικός διάλογος λοιπόν θα πρέπει να γίνεται και να έχουμε αύξηση αύξηση, πιο, πιο, πιο συχνότητα συναντήσεων μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους εκπροσώπους της. Άρα, περισσότερες αντίσεις σημαίνουν περισσότερο συντονισμό, περισσότερη ελοκατανόηση. Και έτσι θα καταλάβουμε καλύτερα το τι πάει να πει επικουρικότητα και τι πάει να πει αναλογικότητα. Ένα από τα προβλήματα τα οποία αναδύονται από την συζήτηση είναι η αποκλίνουσα ερμηνεία αυτών των ενιών από πλευράς κάποιων εθνικών κοινοβουλίων. Επομένως, φαίνεται ότι είναι αλήθεια το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμβάθυνε στο θέμα αυτό, προσπάθησε να ε, αναμορφώσει αυτές τις ε, έννοιες. Υπήρχαν και κάποιες ε, εκθέσεις αξιολογικές και νομίζω ότι θα πρέπει τα κριτήρια να τα είχαν ακολουθήσει όλα τα θεσμικό κατά το οποίο δεν έγινε. Οπότε γι' αυτό και έχουμε αποκλίνουσες ερμηνείε και έχουμε διαφορετικές γνώμες και γνωμοδοτήσεις. Αυτό όμως είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να θυγεί στο κείμενό μας γιατί αυτές οι δύο αρχές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν. Και τώρα κάτι άλλο, κάτι άλλο το οποίο δεν έχει αναφερθεί στο κείμενο. Κάτι όμως το οποίο πρέπει να αναδειχθεί. Πρόκειται για ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων. Τι κάνουν σε σχέση με αυτά, ε, αυτές τις δύο αρχές. Το 2012 Περισσότερες μισές ε, γνωμοδοτήσεις αφορούσαν αποκλειστικά την ε, νομοθεσία. Αλλά τα υπόλοιπα όμως ήταν μη νομοθετικές πράξεις. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθούμε σε αυτές τις μη νομοθετικές πράξεις που θα γίνουν όμως οδηγίες, θα γίνουν νομοθετικά κείμενα. Άρα θα πρέπει τα Εθνικά Κοινοβούλια να αποφανθούν τελικά και για τις μη νομοθετικές πράξεις. Και γι' αυτό ακριβώς και αυτό που προσπαθούμε να τονίσουμε είναι αυτό το μέσο, αυτό το είδος τη, την κίτρινη κάρτα. Κάτι που ξεκίνησε το 2012. Δεν το λέμε αυτό στην έκθεση. Όμως το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε ε, για αυτή, την κάρτα για κάποιε εκθέσεις, κάποια κείμενα που στα οποία διαφωνούν στο Κοινοβούλιο. Και τότε λοιπόν ε, επικαλέστηκα ε, την, αρχή με και αναλογικότητα, αλλά κρίθηκε ότι τελικά αυτές οι αρχές δεν είχαν παραβιαστεί. Γι' αυτό σας λέω ότι στο τέταρτο σημείο, στην τέταρτη παράγραφο, μιλά για την κίτρινη κάρτα το κείμενο μας. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά δεν αναγνώρισε αυτό τον θεσμό, αυτό το μέσον της μη αιτιολογημένης γνώμης. Το 2014 επίσης χρησιμοποιήθηκε αυτή η κίτρινη κάρτα για πολλωστή φορά και για πολλωστή φορά πάλι δεν αναγνώρισε την μη αιτιολογημένη γνώμη ως θεσμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είπε ότι αφορά ε, κάποιο νομοθέτημα για το οποίο το οποίο παραβίαζε την επικουρικότητα οπότε γι' αυτό και είπαμε ότι τελικά είχαμε την πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οπότε είπαμε ότι με αυτή την κάρτα συμπληρώνεται η γνωμοδότηση. Χρειάζεται εξήγηση του πώς λειτουργεί και θα, επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει καλύτερα. Στο σημείο 5 μετά μιλούμε ε, για την αρχή think small first. Δηλαδή, ε, το πούμε αλλιώ, θα πρέπει κανείς να σκέφτεται στα πλαίσια παγκοσμιοποίηση και να ενεργεί τοπικά. Άρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα εμπλέκονται σε τοπικό επίπεδο ε, οι επιχειρήσεις. Και έτσι θα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες των πολιτών. Να εκμεταλλευτούμε επομένως κάθε τρόπο ε, δικτύωσης. Ευχαριστούμε ακούσουμε τη Γιούτα Στάινρουκ για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστούμε. Δυστυχώς ε, η συνάδελφος κυρία Ρέγνερ έχει ένα πολύ σημαντικό ραντεβού και δεν μπορεί να... Δεν μπορούσε να συμμετάσχει στη συζήτηση. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Είναι πολύ καλή η βάση για τις μελλοντικέ μας εργασίες. Ε, μέσα στην έκθεση αναφέρονται 88 ε, αιτήσει των Εθνικών Κοινοβουλίων για τήρηση της αρχής επικουρικότητας. Ε, προσφυγή λοιπόν στη διαδικασία της κίτρινης κάρτας. Το θέμα είναι αν τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν τους απαιτούμενους πόρους για να παρακολουθούν το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κάνει ό,τι θα έπρεπε για να ασκήσουν τα Εθνικά Κοινοβούλια τον ελεκτικό τους ρόλο. Οι σοσιαλιστές ε, θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ θετικό όταν ε, τα εθνικά κοινοβούλια εξετάζουν υπό το πρίσμα της ε, επικουρικότητας μια έκθεση. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε αυτή τη δυναμική διαδικασία δυναμική νομοθετική διαδικασία για να αποφεύγουμε και τα περιτά νομοθετήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά θα προσπαθήσουμε με τροπολογίες να εμπλωτίσουμε αυτή την έκθεση και ελπιστούμε ότι θα καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τώρα η κυρία Χέλγα Στίβενς για να κάνει κάποιες ε, τελικές παρατηρήσεις και να κλείσει και αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η κυρία Στίβενς, σας ευχαριστώ. Με ενδιαφέρον άκουσα και τις δύο πλευρές και όλα τα σχόλια και θα τα περιλάβω όσο μπορώ. Επίσης, με την ε, αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή θα επανέλθουμε μετά τις διακοπές του Πάσχα. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να τα συζητήσουμε τα πράγματα αυτά. Υπάρχουν ίσως κάποιες ελλείψεις στο σχέδιο εκθέσεως. Έχουμε κάποιους περιορισμούς βέβαια λόγω του αριθμού των λέξεων που επιτρέπονται. Θα θέλαμε να προσθέσουμε πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά αναγκαστικά θα περιοριστούμε στα πιο ουσιώδη. Τα σχόλιά σας πάντως είναι ιδιαίτερα καλοδεχόμενα. Το σχέδιο μπορεί να περιλάβει και τις γνώμες αυτές. Απομένως θα, τις, θα κάνω προσπάθεια να τις περιλάβουμε. Ευχαριστώ πολύ που μου τις θέσατε υπόψη. Σας ευχαριστώ. Προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών 17 Τετάρτου το μεσημέρι. Ψήφος εδώ στις 28 Μαΐου και 16 έως 17 Ιουνίου η επόμενη φάση τελευταία. Και τώρα έρχομαι στο υπαριθμόν 12 της ημερησίας διατάξεως Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών μετά το 2015. 112 τροπολογίες επί του σχεδίου γνωμοδοτήσεως. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κασλόφσκα Ρατζιεβίτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι αληθές ότι η γνωμοδότησή μου έχει ε, υποβληθεί και έχει συγκεντρώσει ήδη 112 τροπολογίες. Ευχαριστώ όλες και όλους που κατέθεσαν τροπολογίες, οι οποίες τροπολογίες πιστεύω ότι θα καταστήσουν την ε, αντιμετώπιση του προβλήματος καλύτερη βελτιώνουν την ποιότητα του κειμένου. Είμαι ικανοποιημένη που μάλιστα μπορώ να υπερβώ το όριο των 200 λέξεων που είχε επιβληθεί στο αρχικό κείμενο. Μέχρι τώρα μπόρεσα να καταλήξω σε 12 συμβαστικές τροπολογίες. Ακόμα τώρα επεξεργάζομαι το κείμενο της γνωμοδοτήσεως και έως τώρα έχω διατηρήσει εντονότατη αλληλογραφία με ε, τους ε, άλλους ε, σκιώδης και πολύ καλά τα έχουμε πάει με πολύ καρποφόρο συνεργασία. Μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ικανοποιητικές διατυπώσεις, ικανοποιητικές για όλα τα μέρη, που σημαίνει ότι βελτιώνεται και η ποιότητα των τροπολογιών. Η συζήτηση τώρα περιστρέφεται γύρω από τον ρόλο ανδρών και γυναικών και διευκολύνσεις για τους γονείς αλλά και για τους ηλικιωμένους και ασθενείς, όχι μόνο για τα παιδιά. Επίσης ε, εύκαμπτα ωράρια εργασίας τις ε, γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, την απόσταση των αμοιβών ανδρών και γυναικών και ούτε καθεξής. Επίσης την ε, συμμετοχή των μητέρων στην αγορά εργασίας, κάτι που θεωρώ σημαντικό και θα δώσουμε και συνέχεια. Αναφέρω και την οδηγία για την άδεια μητρότητας και για τη γονική άδεια και την άδεια πατρότητας ζητούμε εμείς την εφαρμογή της ε, οδηγίας που είχε ψηφίσει η κυρία Ρέντινγκ, που είχε προωθήσει η κυρία Ρέντινγκ, για τη συμμετοχή γυναικών ε, στα ε, διοικητικά συμβούλια εισηγμένων στα χρηματιστήρια εταίρειων, καθώς και μιλούμε και για το πρόβλημα πολλαπλών διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Το ίδιο και για το mobbing, ε, σεξουαλική παρενόχληση στον τόπο εργασία και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι όλες και όλους για τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει. Ελπίζω το κείμενό μου να συγκεντρώσει σημαντική πλειοψηφία. Ευχαριστώ κύριε Γκέρικε. Είστε σκιώδης σύγητης. Δεν έχει ούτω. Δεν το γνωρίζετε κύριε Γκέρικε. Δεν υποχρεούστε να πείτε τίποτε αν δεν θέλετε. Ναι, μιλούσαμε με την κυρία Κοσλόφσκα και ήδη αναφέρθηκε στις τρομολογίες μου. Κοιτάξτε, μιλούμε για για τα θήλαια ας πούμε γενικά δηλαδή και οι μητέρες θήλαια είναι που έχουν φέρουν βεβαίως μια ιδιαίτερη ευθύνη για την κοινωνία και πρέπει επομένω να μπει ξεχωριστά. Ε, αυτό, αρκούμε σε αυτό για την ώρα. Α, η κυρία Αρενά που εκπροσωπεί την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ε, ξέρω ότι έχουν καταδεθεί πολλές τροπολογίες και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Με λίγες διαφωνίες διαφωνούμε κάθετα, αντίθετα. Θα θέλαμε ε, να συμπεριληφθούν κάποια σημαντικά ζητήματα μέσα, ε, μέσω των τροπολογιών. Η κατάσταση, παραδείγματο χάρη, ε, που να απέχει από το στόχο μας για την ισότητα των δύο φύλων. Δεύτερον, λαμβάνεται υπόψη αυτό στη στρατηγική 2020 και ε, στην άσκηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το, ε, κυρίως για να επιτύχουμε και τους στόχους μας ε, για την απασχόληση 75% για τις γυναίκες και λιγότερο από 20 εκατομμύρια όχι μόνο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και οικονομικής αποτελεσματικότητας. Ε, το τρίτο ζήτημα είναι η διάκριση κατά των γυναικών ως προς την απασχόληση στα ε, κάθετα, ως προς τα κάθετα και τα εγκάρσια ζητήματα. διάκριση κατά των γυναικών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, κυρίως όταν πρόκειται για πολλαπλές ε, διακρίσεις, ε, χρώμα του δέρματος, ε, αναπηρία, τόπος καταγωγής, πέρα δηλαδή από το ότι είναι κάποιος γυναίκα μπορεί να υφίσταται διακριτική μεταχείριση για μια σειρά από λόγους. Επίσης, ε, επενδύσεις ε, στους, ε, στις υποδομές φύλαξης των παιδιών για να εκπληρωθούν οι στόχοι της Βαρκελόνης. Επίσης, γονεακή άδεια, μητρική πατρική άδεια για να προωθηθεί η απασχόληση των γονεών, Επίσης, συμφιλίωση οικογενειακής και επιχειρηματικής επαγγελματικής ζωής, καλύτερος επιμερισμός των καθηκόντων στο σπίτι και ούτω κάθε Υπάρχει και κάτι για το οποίο η συγκήτρια δεν έχει ε, εισηγηθεί κάποιο συμβασμό και καταλαβαίνω γιατί ε, θέλει να καταψηφίσει την τροπολογία μας υπαριθμών 78 για την ε, στρατολόγηση των γυναικών που επιθυμούν να υπάρχει αντιστροφή του βάρους απόδειξης όταν υφίστανται μία απόρριψη στην διαδικασία πρόσληψης Ξέρετε, όταν υπάρχει διακριτική μεταχείριση είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αντιστροφή του βάρους απόδειξης. Ε, γι' αυτό καταθέσαμε αυτή την τροπολογία. Τέλος, υπάρχουν ε, τροπολογίες σε σχέση με τις μη παραδοσιακές ε, σεξουαλικές ταυτότητες και τις, διακρι... μορφές διακριτικής μεταχείρισης που μπορεί αυτό να επισύρει δεν έχουν γίνει ε, κατά τη γνώμη μου αρκετά πράγματα για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπρόσθετες μορφές διακριτικής μεταχείρισης. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ η συγγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Θα ήθελα κι εγώ να σας ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι έχω λάβει υπόψη τα περισσότερα από αυτά τα σχόλια, όμως ε, σε σχέση με αυτά που μας είπε η τελευταία συνάδελφος, δύσκολα μπορεί κάποιος ε, να καταλήξει σε ένα κείμενο που θα τύχει ε, καθολικής αποδοχής. Ε, αποσκοπούμε μόνο σε μια πλειοψηφική αποδοχή του κειμένου. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε και πολύ λυπούμε που τα θέματα ισότητας των δύο φύλων πάντοτε καταλήγουν στο τέλος της μερίσιας διάταξης όταν έχουμε πραγματευτεί τα σε εισαγωγικά σοβαρά ζητήματα. Θα φροντίσουμε όμως να μην συμβεί αυτό ξανά συχνά στο μέλλον. Στις 16 Απριλίου θα ε, ψηφίσουμε για την έκθεση εδώ τότε δηλαδή που θα συνεδριάσουμε και την επόμενη φορά στις 9 μέχρι τις 6.30 στις Βρυξέλλες. Τελειώσαμε νωρίτερα. Και θα έχουμε και μία ολιγοήμερη διακοπή, ή μάλλον πάνω από μία εβδομάδα. Σας ευχαριστώ όλους. Για τη σκληρή μας δουλειά με την ψηφοφορία τα καταφέραμε όμως με πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ και παρόλα αυτά δεν έκλεισε ούτε και η φωνή μου. Ευχαριστώ.